Meine Κυρίες και κύριοι, περνάμε τώρα στην έκθεση Γιαννάκου. Σχέδιο έκθεση, έκθεσης για τις ε, στρατιωτικές δομές της Ένωσης. Κύριε Λάμστορφ, κύριε Πρόεδρε, πριν πάμε στην ψηφοφορία, θα ήθελα να κάνω μια πρόταση ναι, βεβαίω, αλλά να κάνω πρώτα την εισαγωγή μου. Δεν έχει σχέση με την ψηφοφορία, λέει ο κύριο Λάμσδορφ. Θέλω να επανέλθω στη συζήτηση για το Ιράκ χτε στην Επιτροπή μα. Θα πρότεινα τέτοιε συζητήσει στο μέλλον να γίνονται κατά τρόπον που θα επιτρέπει να μην ε, ε, μονοπολούν τη συζήτηση συνάδελφοι οι οποίοι δεν είναι ούτε τακτικά ούτε αναπληρωματικά μέλη και εμφανίζονται μόνο για κάτι τέτοια ερωτήματα αυτό το οποίο, δεν μου αρέσει να λέω τις λέξεις, αλλά αυτό το οποίο συνέβη χτες ήταν αναξιοπρεπές για το Κοινοβούλιο. Θα μπορούσε ίσως η γραμματεία να σκεφτεί πώς μπορούμε να αποφύγουμε τέτοια πράγματα στο μέλλον, γιατί πάρα πολλοί συνάδελφοι χτες ήταν οργισμένοι για αυτό το οποίο συνέβη. Και εν μέρη συμφωνώ και εγώ. Ευχαριστώ κύριε Λάμσδορφ. Θα το συζητήσουμε στο Προεδρείο αλλά δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα αλλάξει κάτι. Από όλους τους ομιλητές ε, τους χρησινους δυο δύο-τρεις δεν ήταν μέλη της Επιτροπής. Γιατί και εγώ είδα τον κατάλογο τελικά ποιοι ήταν μέλη και ποιοι όχι, γιατί είχα και εγώ αυτή την αίσθηση. Α, το το δεύτερο τώρα, ποιοι έρχονται εδώ πέρα, αυτό είναι ζήτημα των ε, συντονιστών. Δεν θα εμπλακώ εγώ ως πρόεδρος, δεν μπορεί να είναι δουλειά μου ε, να ψάχνω για ποιο λόγο μιλάει ο καθένας. Ε, πρέπει και άλλοι να, να μπορούν να μιλάνε. Αν έρχονται οργανωμένοι είναι και αυτό πολιτικό τους δικαίωμα. Ε, Βεβαίω, εντάξει, δεν μπορεί να μου άρεσε, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορώ και να το εμποδίσω. Έτσι, για να το πω χήμα. Αλλά θα το συζητήσουμε στο διευρυμένο Προεδρείο, αν έχει κανείς κάποια ιδέα. Εγώ προσωπικά πρέπει να πω πως πραγματικά απορώ. Δηλαδή, Να σκεφτούμε παραδείγματος χάρη τι, τι θα γινόταν στην χώρα μας αν υπήρχε μια περιοχή 30 τετραγωνικών χιλιόμετρων την οποία την διεκούσαν μόνο παράνομοι ε, αλλοδαποί. Σκεφτείτε δηλαδή τι γίνεται με αυτούς τους ε, καταβλισμούς. Στο Άστραφ. Ε, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι τέτοιο. Ε, Υπάρχουν τέτοιε καταστάσει, υπήρξαν τέτοιε καταστάσει στη Νότια Αμερική, στη Χιλή και πάλι δεν είναι πλήρω συγκρίσιμε. Και θα πρέπει να δούμε, όπω είπα, αν ισχύουν τέτοια πράγματα. Αν ισχύουν είναι πραγματικά ένα δραματικό σκάνδαλο. Και μετά, σκε... σκεφτείτε, κάθε στιγμή, ε, Επίση σκεφτείτε το εξή, κάθε Ιρακινός αυτή τη στιγμή κινδυνεύει πολύ περισσότερο από τους ανθρώπους σε αυτό το στρατόπεδο και είναι πραγματικά ε, τελείως δυσανάλογο αυτό το οποίο έγινε. Όταν δεν είχε λάβει χώρα η επίθεση αυτή είχαμε περάσει πράγμα το ψήφισμα για την προστασία των ανθρώπων. Αλλά εντάξει τώρα πολιτικά δεν μπορώ να, να συμφωνήσω με αυτά τα οποία έγιναν έτσι και νομίζω πως ο κύριος Κόμπλερ εκεί πέρα έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και θα ήθελα πραγματικά να γραφτεί αυτή η φράση στα πρακτικά. Και πραγματικά πρέπει να το συζητήσουμε ότι ήταν ε, τελείως ε, μη ισορροπημένη η κατάσταση και πρέπει να το πούμε. Ε, γι' αυτό και εγώ θα συνεχίσω να στηρίζω τον ε, κύριο Κόμπλερ ε. και νομίζω πως αυτό εκπροσωπεί και την πλειοψηφία της Επιτροπής. Και θα συνεχίσω να το κάνω και να το λέω και δημοσίως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα, συμφωνώ πλήρως μαζί σας. Θα το συζητήσουμε στο διευρυμένο Προεδρείο. Θα ήθελα να πω μια που, δεν τα ακούσατε ίσως μια που η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει 12 εκατομμύρια ευρώ ε, δικά μας λεφτά, μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Λέδη Άστον ή τις υπηρεσίες της να έρθουν εδώ πέρα να τη ρωτήσουμε πού πάνε τα λεφτά αυτά και να βοηθήσουμε να επαναγκατασταθούν ε, οι άνθρωποι που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να πάνε αλλού και υφίστανται αυτή την πλήση εγκεφάλου και την παρενόχληση και την στέρηση της ελευθερίας ε, που αναφέρθηκε χθε. Και επί τη ευκαιρία, οι επιθέσεις δεν είναι μόνο εναντίον του κυρίου Κόμπλερ, αλλά και κατά της ε, Ντάνα Ιμπάσκοβα, της επικεφαλής αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι μέλος αντιπροσωπείας και είμαι από τα λίγα μέλη ε, που πηγαίνουν εκεί πέρα, πέραν από αυτούς που υποστηρίζουν τη Μουτζαχεντίν του λαού. Και πραγματικά ε, δεν είναι σωστό αυτό το οποίο συνέβη με την προσωπική επίθεση των κύριο Κόμπλερ και την ε, κυρία Γιάννα Ιμπάσκοβα και εγώ διαμαρτυρήθηκα. Πραγματικά καταστρέφεται έτσι η επιρροή μας στο Ιράκ και η δυνατότητά μας να έχουμε σχέσεις με τους Ιρακινούς συναδέλφους. Ε, έρχονταν πολύ πιο συχνά, τώρα δεν έρχονται, γιατί δεν έχει νόημα. Συζητάμε συνεχώς για το θέμα αυτό, τους Μουτζαχιντίν του λαού. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω λίγο. Μια που μιλάμε για πρόσφυγες και τη κατάστασή τους, πρέπει να θυμόμαστε πως κάποιοι από αυτούς έχουν μετεγκατασταθεί σε νεκροταφεία μετά από τις επιθέσεις στο Άσραφ όχι μόνο από Ιρακινούς αλλά και από φρουρούς επανάστασης από το Ιράν που μπαίνουν σε άλλη χώρα με τη στήριξη της Ιρακινής κυβέρνησης μετά μιλάμε για πρόσφυγες ως Μουτζαχεντίν και υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων ε, νεκρών, ε, τραυματιών ε, που είναι γεννημένοι στο Ιράκ. Δεν είναι ξένοι Μουτζαχεντίν. Αυτά για την τωρινή συζήτηση. Και για τον κύριο Κόμπλερ. Εγώ τον ρώτησα δύο πράγματα χθες. Πρώτον, ένα γενικότερο και πρακτικό για την έρευνα διερεύνηση των κατηγοριών και το επόμενο αφορούσε την παρέμβαση του Ιράν στο θέμα και τη συνεργασία του με την Τεχεράνη. Ε, δεν απάντησε σε καμία ερώτηση, οπότε ε, δεν θα υπερψηφίσω εγώ. Danke. Κυρία Λούνατσεκ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να αποσαφηνίσω εξ ονόματο τη ομάδα μου ότι υποστηρίζω πλήρω ε, την παρατήρηση που έκανε ο πρόεδρο Μπρόκ εδώ. Και ακόμα και στο διευρυμένο Προεδρείο να συζητηθεί απόψε. Και εξ ονόματο τη ομάδα μου θα, θα υποστήριζα το να αποσταλεί μια επιστολή προ τον κύριο Κόβλε. Σα ευχαριστούμε θερμά λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα άτομα υποστηριζόντουσαν παλαιότερα από τους κομμουνιστές όταν υπήρχε αυτή η κατάσταση σε σχέση με το Ιράν. Με εκπλήσει η τροποποίηση υποστήριξη σε ένα κύμα ανακύκλωσης που απορρέει σε αυτό το σώμα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι, αυτά μου δημιουργεί κάποια σύγχυση, ας το πω έτσι, αυτό. Και περνάμε τώρα στο θέμα της κυρίας Μαριέτας Γιαννάκου. Η έκθεση αυτή δεν μου δημιουργεί σύγχυση. Θέλετε να προσθέσετε κάτι κυρία Γιαννάκου. Κύριε Πρόεδρε, έχω στείλει από χθες και την ε, λίστα ψηφοφορίας ε, όπως την προτείνω εγώ ε, και όλα τα σχετικά εδώ και μέρες. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι γνωρίζουν και τις προφορικές τροπολογίες, τα πάντα και νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ και περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 22 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 23 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 24 με προφορική τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 25 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 26 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 31 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 34 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 35 και 36 υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν 37 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 38 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 39 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 40 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 41 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 42 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 43 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 44 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 46 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 47 υπέρ κατά αποχές 47 υπέρ και πάλι κατά αποχές εγκρίθηκε να ελέγξουμε λέτε ωραία 47 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται δεν έχω την κάρτα μου όμως εγώ άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ ναι, αλλά δεν έκλεισε η ψηφοφορία, μπορώ να ψηφίσω ακόμα. Μάλιστα. Τώρα πέρας ψηφοφορίας, έκλεισε η ψηφοφορία. Με 24 ψήφους υπέρ 18 εναντίον εγκρίθηκε. 48 τώρα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 49 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 50 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Συμβασμός 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 53 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπο, τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 64 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 65 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 66 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 67 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. 68 υπέρ, κατά απόχέ, απορρίφθηκε. 69 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 72 υπέρ κατά αποχές εγκρι... απορρίφθηκε 73 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 74 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 75 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 77 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 78 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 79 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 80 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 81 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 83 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 84 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 85 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε προφορική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 87 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 90 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 95 με προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 97 και 98 υπέρ αυτών κατά αποχές απορρίφθηκαν. 99 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 100 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 101 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 102 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 104 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 1 με προφορική τροποποίηση 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δύο υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σύνολο του έργου. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα 33 ψήφοι υπέρ, 11 εναντίον. Εγκρίθηκε. Θερμά συγχαρητήρια στην κυρία Γιαννάκου. Πάμε τώρα στην έκθεση. Εσείς τι λέτε παρακαλώ. Yeah, bitte ναι, παρακαλώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, απλώς ήθελα να πω ότι σε αυτό το θέμα η ομάδα μας καταθέτει minority report και για να μην επανέλθω, αναφέρω ότι και στο επόμενο θέμα καταθέτουμε επίσης Minority Report. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίω έχετε το δικαίωμα. Έχετε το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ για να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους με τους οποίους ε, συνεργάστηκα και πραγματικά έκαναν ουσιαστικέ ε, συνεισφορές και ιδιαίτερα τον βοηθό μου τον Αλέξανδρο Περέιρα που συνεργάστηκε και εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά. Οπότε, Περνάμε στην ε, συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 45 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Μετά τροπολογία 48 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 49 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 50 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Τι ήτανε, τι συνέβη με την 55. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Όχι. 63 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 73 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 78 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 79 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 80 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 81 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 82 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 83 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 19 εναντί 24. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Προφορική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 88 υπέρ. Κατά. Νομίζω γίνεται δεκτή. Να την επαληθεύσουμε. Νομίζω ότι... Πέρας. Απορρίπτεται. 21-23. Ποια ήταν αυτή. Μάλιστα. 89 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην 94. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 95 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ορίστε. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές δεκτή 112 ηλεκτρονική ψηφοφορία πέρας 27 υπέρ, 17 κατά. Δεκτή. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. 113, ε. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεν μπόρεσαν οι πράσινο-δεξιοί να επιβληθούν. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 119 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά αποχές η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δεύτερη απόπειρα. Πέρας. Με δύο ψήφους διαφορά. Δεκτή. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Προφορική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην προφορική τροπολογία 7. Υπέρ. Προφορική τροπολογία 7. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 128 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. αποχέ, Δεκτή. μερο δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Προφορική τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 139 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 141 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική ψηφοφορία. 141. Πέρας. Μάλιστα. Δεκτή. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 144 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβεστική 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 146 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. 34 με 10, αλλά παρακαλώ να ε, σηκώνετε τα χέρια σας άλλη φορά. Ναι, ναι. Πιείτε καφεδάκι. Ορίστε. 149 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 157 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 159 υπέρ, κατά αποχές Απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ. Κατά αποχές Ξανά 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Τώρα ε, είστε υπέρ κατά ή ε, αποχή. Τι. Μα είχατε ακόμα το χέρι σηκωμένο. Δε, τα πάντα ψηφίσατε. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία. Όχι, λάθος. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μετά 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 κατά πίπτη 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή προφορική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3 και 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 έως 8 μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί 5 έως 8 υπέρ κατά αποχές δεκτές 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή η κοινωνική ψηφοφορία στο σύνολο Με το ίδιο αποτέλεσμα όπως και η προηγούμενη έκθεση. Α, όχι, όχι και μία αποχή. 33 υπέρ, 11 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια για Νέτα. Μαριέτα. Ε, Άννα, Μαριέτα. Άννα, ναι, συγγνώμη. Ε, για δώσε, δώσε. Συγγνώμη. Δώσε, Äh, Περνάμε τώρα στην έκθεση του Κόμιτα, του Κόμι Λάμστορφ. Θέλετε να πείτε κάτι, παρακαλώ. <clears throat> Θέλω να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές ε, και όλους για την καλή συνεργασία. Ωραία, συμβιβασμός 1, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίθηκε. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 25 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 27 υπέρ κατά ασαφές το αποτέλεσμα. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Να. Πέρας ψηφοφορίας. Με 13 ψήφους υπέρ 31 ψήφους εναντίον απορρίφθηκε. απορρίφθηκε. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε περνάμε στην τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 36 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 38 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 41 υπέρ. Κατά. Α, εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε λοιπόν. Εγκρίθηκε. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 45 υπέρ ναι εσείς τι λέτε για πως αποσαφήνιση στην 44 υπήρχε προφορική τροποποίηση ψηφίστηκε και αυτή η τροποποίηση θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό σαφέσα ε? 44 είπα, αλλά όπως έχουμε εδώ έχουμε και την προφορική τροποποίηση. Ισχύει όπως τον κατάλογο ψηφοφορίας. Επειδή θέλω να κάνουμε πιο γρήγορα την ψηφοφορία, δεν διάβασα τα πάντα. Αλλά ψηφίζουμε αυτά τα οποία αναφέρονται στον κατάλογο ψηφοφορίας για τις τροπολογίες πάντα. Με την προφορική τροποποίηση ένα λοιπόν εδώ. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 45 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 46 υπέρ, κατά, αποχές, ασαφές το αποτέλεσμα, ψηφίζουμε και πάλι 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε, εγκρίθηκε, μάλιστα εγκρίθηκε. Πίστεψέ με Μαριέτα, Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία ηλεκτρονικά τώρα, επ' αυτής. 20-19, το είπα, εγκρίθηκε. Μάλιστα. ΔΕΒΕ 12, υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 48 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 49 υπέρ κατά αποχές ασαφές το αποτέλεσμα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχεται πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα 21 ψήφοι υπέρ 18 εναντίον εγκρίθηκε 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε με την ίδια πλειοψηφία 51 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε συμβιβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε Τροπολογία 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στην τροπολογία 58. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε τώρα στην 74, δεύτερο τμήμα της 74, υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Πάμε μετά στην τροπολογία 76, υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 78 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 79 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε 80 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 81 υπέρ όχι σε δύο τμήματα είναι πρώτο τμήμα υπέρ έτσι ωραία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα στις 81 ποιοι είναι κατά ποιοι είναι κατά κατά είπα λέει ο πρόεδρος υπέρ Να προσέχετε λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ. Για το δεύτερο τμήμα λέμε υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 82 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Απορρίφθηκε λέει. Ναι, οι σοσιαλιστές υπερψήφισαν όμως ψήφισαν υπέρ, όχι. Όχι λέγεται από τον συνάδελφο. Ναι, 85 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 86 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 87 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 88 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 88 και πάλι υπέρ κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Να ελέγξουμε και σε αυτή την περίπτωση αποφασίζουν οι φιλελεύθεροι αν θα γίνει δεκτή ή όχι. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα Κάποιοι κομμουνιστές πρέπει να ψήφισαν μαζί με το ΕΛΚ από ό,τι φαίνεται. Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο. Ε, τότε θα πρέπει να καταψηφίσουμε γιατί δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε. Ξαναψηφίζουμε λοιπόν για άλλη μία φορά την 88, εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας. Και αποτέλεσμα, μάλιστα. Βλέπετε ποια είναι η μεγάλη δύναμη ατομικά του κάθε Ευρωβουλευτή. 89 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. και πάλι βρίσκεται στη, στον κρεμό αυτή. Πέρα ψηφοφορία τώρα. Απορρίφθηκε. 91 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. 92 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 90 93 κατά πίπτη Συμβιβασμός 8 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 96 τώρα. Υπέρ τη 96. Κατά αποχέ απορρίφθηκε. 97 υπέρ. Κατά αποχέ απορρίφθηκε. 98 υπέρ. Κατά αποχέ. ασαφές το αποτέλεσμα. Θα ψηφίσουμε και πάλι. 98 ηλεκτρονικά αυτή τη φορά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Μάλιστα. 22-22 ισοψηφία απορρίφθηκε. Κύριε Παλέτσκης, δεν θα συμμετάσχουμε σε περαιτέρω ύπνο ή λίθαργο. 99 τώρα, μάλιστα. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 100 τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Το ΕΛΚ μόνο του, δεν είδα κανέναν άλλον. ΔΕΒΕ 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. ΔΕΒΕ 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 101 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 102 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. ΔΕΒΕ 1 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. ΔΕΒΕ 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεβε 3 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Δεβε 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Ή πως ψήφισαν οι σοσιαλίστες εκτός από την άλλα. Όχι. Απορρίφθηκε. Οι υπόλοιποι δεν συμμετείχαν. Εντάξει, 103 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεβε 5 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Δεβ 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεβ 8 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Συμβασμός 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Πάμε στην τροπολογία 108 υπέρ κατά 9 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 12 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 15 κατά Κύριε Παλέτσκης, κατά, τι γίνεται. Die Abstimmung ist geschlossen. Πέρας ψηφοφορίας λοιπόν, μάλιστα. 24 ψήφοι υπέρ, 16 εναντίον, εγκρίθηκε. Το ΕΛΚ και η ΓΚΟΕ, συνασπισμός ανίκητος. Μάλιστα, 16 υπέρ, κατά αποχές απορρίφθηκε. 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίθηκε. 1 και 7 υπέρ αυτών κατά αποχές εγκρίθηκαν. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 8 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίθηκε. Και περνάμε τώρα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία στο σύνολο της έκθεσης. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. 38 ψήφοι υπέρ. 6 εναντίον. Εγκρίθηκε. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν. Κόμι Λάμστορφ.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 και σύσταση σε Συμβούλιο Κομισιόν και Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να υπενθυμίσω πως ακριβώς 10.30 θα ξεκινήσει η συζήτηση με την Υπουργό Εξωτερικών του Μπαγκλαντές. Και να υπενθυμίσω στους ε, ε βοηθούς εδώ πέρα πως ε, υπάρχει αρκετά μεγάλη προσέλευση σε τέτοιες περιπτώσεις. Και καλό είναι να υπάρχει γιατί καλό είναι να μην μιλάνε τέτοιοι άνθρωποι απέναντι σε άδεια έδρανα. Παρακαλώ λίγο εκεί οι βοηθοί των σοσιαλιστών να ακούσουν λίγο τον πρόεδρο. Μπα, δεν βλέπω να τους κάνω καμία εντύπωση. Κύριε Παλέτσκης, λοιπόν. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα τελευταία 19 χρόνια το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε 37 ψηφίσματα συγκεκριμένα για τη Λευκορωσία. και μαζί με άλλα κράτη συζητήσαμε 71 φορές την κατάσταση στη χώρα αυτή. Όμως είναι η πρώτη φορά που επιτέλους θα συζητήσουμε για τη Λευκορωσία και τι σχέσει της με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το φω όχι μια αντίδραση στις νέες εξελίξεις στη χώρα αυτή, αλλά προσπαθώντας να αναλύσουμε την κατάσταση και να προτείνουμε συγκεκριμένη πολιτική δράση. Στα μέσα Μαΐου πέρασα τέσσερις μέρες στο Μίνσκ σε επίσκεψη, όπου είχα συναντήσεις με κυβερνητικούς εκπροσώπους και επίσης πολλέ συναντήσεις με εκπροσώπου της Κοινωνία των πολιτών, του εκπροσώπου της αντιπολίτευσης, εμπειρογνώμονε και πρέσβεις ε, στη χώρα. Ε, επέστρεψα με την αίσθηση ότι μπορεί να υπάρχει ευκαιρία να αλλάξουν κάποια πράγματα, να ξαναυπάρξει πολιτικό διάλογο με το Μίνσκ υπό συγκεκριμένε προποθέσει, και αυτό θα είναι ευεργετικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για του πολίτε της Λευκορωσία και θα δημιουργήσει και καλύτερο κλίμα για τι δραστηριότητε των μη κυβερνητικών οργανώσεων, τη αντιπολίτευση και των ελεύθερων μέσων μαζική ενημέρωσης. Αυτή την αίσθηση επιβεβαίωσαν κάποιοι επίσημοι στι Βρυξέλλε, όπου ε, έτσι καλώ σε έξι μήνε θα οργανωθεί μια συνόδος κορυφή για εταιρική σχέση. Βεβαίω υπάρχει η διαταραχή που είχαμε πριν από δυόμιση χρόνια και που είχε χαλάσει την καλή ατμόσφαιρα, αλλά θα χρειαστούν κάποια περαιτέρω βήματα πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι θα απελευθερωθούν πολιτικοί κρατούμενοι και θα αποκατασταθούν στην πολιτική τους δράση. Τα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία ζητούν την ε, επανέναρξη του διαλόγου, του διαλόγου εφόσον βέβαια εκπληρωθούν αυτές οι προϋποθέσεις. Προς στιγμή η επίσημη κυβέρνηση του Μίνσκ στέλνει κάποια μηνύματα προς τις Βρυξέλλες ότι παρά τις δεσμεύσεις της για το ε, πρόγραμμα ε, του Ευρασιατικής Συνεργασίας Υπάρχει μια διάθεση να παρακάμπτουν ε, οι Λευκορώσοι τις ε, υποχρεώσεις τους, ανάλογα με το του συμφέρει προς Ανατολάς ή προς Δυσμάς. Δεν έχει χαθεί όμως τελείως η Λευκορωσία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε μπορούμε και πάλι το αρνητικό κλίμα να το αντιστρέψουμε και να επικεντρωθούμε ε, και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορισμένοι υποστηρίζουν. Αλλά εγώ διαφωνώ με την ε, ιδέα να εγκαταλείψουμε τους Λευκορώσους. Τους 10 εκατομμύρια πολίτες της πρέπει να τους ενισχύσουμε προσπαθώντας να αλλάξουμε τα πράγματα. Διότι περισσότεροι έχουν στενούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι κι αλλιώς από το 2010 ο μεγαλύτερος αριθμός ε, θεωρήσεων Σέγγεν που έχουν ε, εκδοθεί παγκοσμίω εκδίδονται στην Λευκορωσία. Αυτό ο υπολογισμό επιβεβαιώνει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του πληθυσμού τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, α... κρατάει αποστάσει από τη Λευκορωσία, γιατί υπάρχει και ένα οικονομικό πόλεμο σε σχέση με τι θεωρήσει. Είναι πολύ ακριβό το τίμημα των 60 ευρώ. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με τα προξενία μα των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Μίνσκ Επίσης, Οι ουρέ φορτηγών κάποιε φορέ ξεπερνούν τα 15 χιλιόμετρα στα σύνορα. Θα πρέπει όλε οι πύλε, τα σημεία ελέγχου και τα σύνορα να ανοίξουν για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να επισκέπτονται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσω και κάποια πράγματα που προέκυψαν από τη μακρά περίοδο του ψυχρού πολέμου. Υπήρξαν αυστηρέ κυρώσει κατά τη Σοβιετική Ένωση και τα κράτη δορυφόρου τη και για διαφορετικούς λόγους. Θα προσπαθήσουμε, θα έπρεπε λοιπόν τον αποκλεισμό των χωρών του Ανατολικού Μπλοκ να τον δούμε και υπό μια άλλη σκοπιά ότι κάποιοι μεταρρυθμιστές σαν τον Κορμπατσόφ και τους διαδόχους του δεν θα είχαν ποτέ καταφέρει τίποτα εάν δεν άλλαζαν τα στερεότυπα του ψυχρού πολέμου. Αυτά όλα αντιστράφησαν επειδή υπήρξαν τακτικέ επαφέ με πολλού ανθρώπου που βρίσκονταν πίσω από το παραπέτασμα με δυτικού. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Αλεξάνδρ Λουκασέγκο στηρίζεται από περίπου 30% των πολιτών της χώρας. 10 έως 15% των Λευκορώσων στηρίζουν την αντιπολίτευση ωστόσο. Και υπάρχει καχυποψία και ε, διαφωνίες μεταξύ τους, αλλά πρόσφατα παρατηρήσαμε ενθαρρυντικά σημάδια ότι υπάρχει διάθεση να ενισχυθούν οι βασικές πολιτικές τους θέσεις. Ήταν δύσκολο να σκεφτούμε πως θα έχουμε μια καλή επικοινωνία με τους Λευκορώσου, αν δεν οργανωθεί μια κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία. Και κυρίως τα νέα που μαθαίνουμε προέρχονται από δημοσιεύματα στον τύπο. Είναι σύνηθες οι ευρωβουλευτέ να μην μπορούν να λάβουν θεωρήσει και να επισκεφθούν τη χώρα. Και εγώ το έχω ζήσει αυτό. Ωστόσο, ελπίζω ότι η προβλεπόμενη επίσκεψη αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στο Μίνσκ θα λάβει χώρα στα μέσα Ιουλίου. Θα είναι η μόνο μόλις η δεύτερη επίσκεψη από το Κοινοβούλιο εκεί μέσα σε μια δεκαετία. Οι συστάσεις λοιπόν αυτές και η συζήτηση σχετικά ε, θα ενισχύσουν ελπίζω και θα αυξήσουν την προσοχή των Ευρωβουλευτών για τα θέματα της Λευκορωσίας. Είναι πολύ σύντομη η σύσταση που έχω συντάξει με κάποια επικριτικά σχόλια και ελπίζω με τους συναδέλφους να συμπληρώσουμε τα υπερχόντα κείμενα, καταδικάζοντα τι αρνητικέ συνθήκε και δίνοντα ε, έμφαση στι προποθέσει που πρέπει να ισχύσουν για να υπάρξει ευρωπαϊκή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάσει τη αρχή κυρίω more for more, περισσότερα για περισσότερα. Στο σχέδιο σύσταση αναφέρω ότι η βελτίωση τη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη προστασία του είναι κάτι που ήδη το παρατηρήσαμε και το καταγράψαμε το 2012. Η διατύπωση αυτή βασίζεται στα στατιστικά στοιχεία του, ε, ε, του Κέντρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που παρακολουθεί τις ε, ε, συλλήψεις που γίνονται για πολιτικά αίτια. Φάνηκε όμως και μέσω της σύστασης και επειδή υπήρχε η ανάγκη να, να το κείμενο ότι, ότι αυτή η κατάσταση δεν καταγράφηκε επαρκώς. Θα πρέπει λοιπόν να παρανέλθουμε στην αρχική έκδοχη του κειμένου. Ίσως να σφάλουμε, αλλά μετά από 9 χρόνια εργασία στην αντιπροσωπεία με τη, για τη σχέση με τη Λευκορωσία, με συνομιλίες με πολιτικούς και ανθρώπους από τη Λευκορωσία, καταλήγουμε στα εξή. Η κατάσταση στη χώρα θα αλλάξει μόνον όταν η κοινωνία αλλάξει. Και αυτό θα γίνει μόνο εάν πολλαπλασιαστούν οι επαφέ μεταξύ των ε, πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Λευκορωσία η ευημερία και η ελεύθερη σκέψη των Λευκορώσων είναι κάτι που θα πρέπει να στηριχθεί. Όχι ο αυτοαποκλεισμό που προωθείται από την κυβέρνηση της Λευκορωσίας. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε την αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες των στοχευμένων ευρωπαϊκών κυρώσεων και το τι αντίκτυπο έχουν στη ζωή των Λευκορώσων. Νομίζω ότι οι κρίσιμες πολιτικές τους δεσμεύσεις μπορούν να αποδώσουν καρπούς. Ο διάλογος για το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης, εφόσον η Λευκορωσία επισήμως πια αναλάβει τις υποχρεώσεις της και ενισχύσει την κοινωνία των πολιτών, μπορεί να περάσει και σε πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Είμαι ευγνώμων στους συναδέλφους του ΕΛΚ, με τους οποίους συνεργάστηκα στενά κατά την προετοιμασία του πρώτου σχεδίου της σύστασης, καθώς και προς την προς ε, εκπροσώπους διαφορετικών Γενικών Διευθύνσεων και τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, αλλά και ε, του Λευκορώσου του ίδιου, εκπροσωπού τη κοινωνία των πολιτών και άλλου ανθρώπου τη χώρα. Ε, σας Σα ευχαριστώ για αυτήν την ε, συζήτηση. Ελπίζω να συμμετάσχουν όλοι ενεργά και να αλλάξει αυτή η πολύ δυσάρεστη κατάσταση για του ανθρώπου τη Λευκορωσία. Ευχαριστώ. Now is Mr. Lizek. Ο κύριος ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματος του κυρίου πρωτασέβιτς. Είναι αυτή τη στιγμή στο Κίεβο. Ε, θα συναντηθεί με τον κύριο Κλέτσικο και μετά και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Οπότε, όπως είπα, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παλέτσκη εξ ονόματος του κύριου πρωτασέβιτς για την έκθεση αλλά ιδιαίτερα για το ότι από την πρώτη στιγμή ενέπλεξε τον κύριο Πορτασέβιτς ε, στην έκθεση αυτή. Βεβαίω υπάρχουν θέματα τώρα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε στην έκθεση, αλλά υπάρχουν και θέματα τα οποία είναι ξεκάθαρα. Σε γενικές γραμμές δεν είμαστε κατά του μελλοντικού διαλόγου με τη Λευκορωσία και τον ΕΚΕΙ και έτσι των οικιαρχών αλλά πρέπει βεβαίως να δούμε τι θα γίνει και με τις ε, ΜΚΟ που γενικά έχουν μια πάρα πολύ αρνητική θέση για το ότι συμβαίνει στην ε, Λευκορωσία και ότι δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη πρόοδος. Οπότε ό κόμματα της αντιπολίτευσης λοιπά, Όλα αυτά δεν υπάρχουν και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα της πολωνικής μειονότητας που δεν έχει λυθεί. Και οι πολωνικές ενώσεις στη Λευκορωσία ε, διώκονται με διάφορους ε, τρόπους και δεν μπορούν να εμπορευθούν ελεύθερα. Βεβαίω υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο εκκρεμεί, οι ελεύθερες εκλογές. που δεν μπορούν να γίνουν και από ό,τι φαίνεται δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι στο προσεχές μέλλον. Οι σχέσεις μας στο μέλλον ε, πρέπει να οδηγηθούν μέσω δίκαιων και ελεύθερων εκλογών, να μπορούν να κατέβουν στις εκλογές ε, εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, να έχουμε εκλογές υπό διεθνή επίβλεψη, να μην υπάρχει νοφία, όλα αυτά δηλαδή που πρέπει να γίνουν σωστά. Επί της αρχής λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε σωστό διάλογο με το κοινοβούλιο γιατί δεν είναι αξιόπιστη εταίρη. Οπότε τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Αλλά όπως είπα δεν έχουν λυθεί ακόμα αυτά τα ζητήματα στη Λευκορωσία, ζητήματα της κοινωνίας των πολιτών, λειτουργίας της αντιπολίτευσης, ε, Υπάρχουν ε, ακόμα πολιτικοί κρατούμενοι στη Λευκορωσία. Και βεβαίως ο κύριος ε, Προτασέβιτς ε, συνεργάζεται στενά με τον κύριο Παλέτσκη, αλλά θεωρούμε πως οποιαδήποτε μορφή διαλόγου πρέπει να γίνει υπό κάποιες βασικές συνθήκες που δεν συντρέχουν. Σας ευχαριστώ, εκπροσωπήσατε πάρα πολύ καλά τον κύριο Πρωτασέβιτς, Κυρία Νέιτς, θέλετε τον λόγο? Όχι. Απουσιάζει ο σκιοδησυγητής, δεν έχουν από τίποτα. Για τους πράσινους, κύριε Σούλτς, έχετε τον λόγο. Ε, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον κύριο Παλέτσκης πολύ εκτεταμένη και πολύ καλή έκθεση και τον ευχαριστώ και για την διάθεση συνεργασίας που επέδειξε, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να μάθουμε. Παραδείγματο χάρη, εμείς εκτιμούμε διαφορετικά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν βλέπουμε καμία βελτίωση, συμφωνούμε με τη Γιάσνα, την Επιτροπή του Ελσίνκη και την Επιτροπή 97, τη Χάρτα 97, μπορούμε να πούμε μάλιστα πως επιδεινώθηκε η κατάσταση, υπάρχουν συλλήψεις, βασανιστήρια, πολιτικοί κρατούμενοι, δημοσιογράφοι και ακτιβιστές διώκονται. Θα αναφέρω εδώ την αυθαίρετη σύλληψη του Αλέξη Μιαλίτσκη που διαπίστωσε κάποια πράγματα. Επίσης, δεν ε, πετράπει στον ειδικό αποσταλμένο του ΟΗΕ να μπει στη χώρα και διάφοροι παρατηρητές του ΟΣΕ τραυματίστηκαν. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα των πολιτικών κρατουμένων. Στο θέμα του εξυγχρονισμού Τώρα τι να σου πω, εγώ το βρίσκω κάτω πολύ αμφιβολό στην περίπτωση της Ρωσίας. Το νόημα δεν είναι να εξυγχρονιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον στην άλλη πλευρά βρίσκεται η αναγκαιότητα εξυγχρονισμού, αλλά δεν βλέπω καμία διάθεση και δεν μπορούμε να μιλάμε για εξυγχρονισμό αν δεν είναι διατεθειμένη για κάτι τέτοιο η άλλη πλευρά. Για τις κυρώσεις προσοχή πρέπει να έρθουν εγκαίρως και να σκεφτούμε γιατί δεν λειτουργούν οι κυρώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά παραθυράκια που χρησιμοποιούνται, οπότε πρέπει να δούμε την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων. Όσον αφορά την διακοινοβουλευτική συνεργασία, δεν ξέρω τι κάνει εδώ πέρα στην έκθεση. Σε ένα ψήφισμα του Δεκεμβρίου είπαμε ξεκάθαρο πως δεν αναγνωρίζουμε το κοινοβούλιο του Μίνσκ, δεν συνεργάζεται στη Euronest, είναι το μοναδικό κοινοβούλιο που δεν εκπροσωπείται στη Euronest και το είπε νομίζω ο συνάδελφος βασικό κριτήριο είναι ελεύθερες και μυστικές εκλογές που μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει. Οπότε κάποια επικοδομητικά πράγματα με τα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε αλλά νομίζω πως ε, πρέπει ξεκάθαρα να αναφέρουμε βεβαίως και τα ελλείμματα. Σας ευχαριστώ ο κύριος Τάνοκ για τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές. Uh, Ακούσα προσεκτικά όσα μόλις είπε ο κύριος Παλέτσκης και σέβομαι ιδιαίτερο στην εντυμότητά του το γεγονός ότι προσπαθεί να συνεισφέρει νέες ιδέες στην όλη συζήτηση. Αλλά με τα λύπης μου να πω ότι Κάποια στιγμή η Λευκορωσία ήταν η κούβα της Ευρώπης, ε, αυτό το λέγαμε πριν μια δεκαετία. Δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει ποτέ, πολύ, ιδίω ω προ την καταπίεση των μέσων μαζική ενημέρωση. Πολλέ πολιτικέ δεσμεύσει εκφράστηκαν, διτυπώθηκαν, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα στην πραγματικότητα. Με τον Λουκασέκο δεν γίνεται τίποτα. Παραμένει ένα παρανοϊκό και ε, απρόβλεπτο δικτάτορα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πραγματικό δίλημα με ισχυρά επιχειρήματα και από τι δύο πλευρέ Δηλαδή να ξεκινήσουμε ένα διάλογο με τη Λευκορωσία ή να τα παρατήσουμε. Συνάντησα τον κύριο Μανκέιβ, ο οποίο ακολουθεί τη γραμμή του κυρίου Παλέτσκη και κάποιου άλλου από την αντιπολίτευση στην Πρατισλάβα. Ήταν δύσκολε οι συζητήσει, γιατί ακόμα και η αντιπολίτευση κατά του Λουκασέγκο είναι πολύ ε, διχασμένη σε σχέση με την προσέγγιση που θα ακολουθήσουν. Η ομάδα μου προ την ισορροπία που αναζητούμε μάλλον είναι υπέρ τη αποχώρησης από τις προσπάθειε σύναψη σχέσεων με τη Λευκορωσία. Δεν υπάρχει πρόοδο σε θέματα δημοκρατία, σε θέματα θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το να αρθούν οι στοχευμένε κυρώσει είναι πρόημο σε αυτό το στάδιο, αλλά βλέπουμε να μην υπάρχει σοβαρό αντίκτυπο στην οικονομία τους, ε, της Λευκορωσίας τόσο ή άλλως θα πρέπει να δούμε και άλλη πρόοδο για να προχωρήσουμε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βλέπουμε ότι η Λευκορωσία παραμένει μια θλιβερή ιστορία, ε, ιδίως για του ε, πολίτε τη χώρα, Πρέπει να δούμε αλλαγέ τα επόμενα δύο χρόνια και να ξεκινήσουμε τουλάχιστον προσπάθειε να είμαστε σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών. Ενδεχομένω να διευκολύνουμε τους λευκορώσου φοιτητέ, επαγγελματίε, με τι ε, θεωρήσεις του να έρθουν προ την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την κυβέρνηση δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά. Πρόεδρο. ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Γκάλερ. Ευχαριστώ. Ήδη πολλά ακούστηκαν. Ε, θέλω να το επαναλάβω. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παλέτσκης για την ε, συνεργασία που που είχαμε. Όλα τα θέματα νομίζω έχουν αναφερθεί. Στο σημείο 1α όπου μιλάμε για ανεφόρον απελευθέρωση των πολιτικών ε, κρατουμένων θα ήθελα και εγώ να το τονίσω και στην εισαγωγή του τώρα έκανε κάποια κριτική αλλά βεβαίω ε, λέει εκεί πέρα πω ναι, υπάρχουν κάποιοι όροι. Δεν ξέρω, ίσω πρέπει να το δούμε κάπως καλύτερα αυτό το ζήτημα για τη βελτίωση των σχέσεων. Δηλαδή, αν υπάρξουν περισσότερες μεταρρυθμίσεις μπορεί να γίνουν περισσότερα πράγματα. Κάποια πράγματα που υποστηρίζω περισσότερο αφορούν τις επαφές με την κοινωνία των πολιτών. Εδώ πέρα πρέπει πραγματικά να προσπαθήσουμε τα τέλη για τη θεώρηση να μειωθούν. Δεν βοηθάει, νομίζω, τις επαφές των ανθρώπων. Και νομίζω πως ε, έτσι θα βοηθήσουμε τον κόσμο και όχι το καθεστώς. Και θα μπορέσουν να μεταφέρουν ε, τις εντυπώσεις τους στη χώρα τους και να διατηρήσουν τις επαφές που έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό και νομίζω κάτι πρέπει να κάνουμε να πιέσουμε και εμείς τη διοίκηση εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούζεκ. Ε, dziękuję bardzo, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ Πρόεδρε θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την προετοιμασία της σύνταξης αυτής της έκθεσης. Ίσως μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις εδώ στην αίθουσα. Συμβαίνει συχνά αυτό, αλλά είναι σημαντικό να συζητάμε ο ένας με τον άλλον ανοιχτά και ειλικρινά και κάθε να εκφράζει ανοιχτά και ειλικρινά τις θέσεις του. Αυτή η έκθεση εμπεριέχει πολλά και από αυτόν τον ανοιχτό ειλικρινό χαρακτήρα. Ανοιχτό χαρακτήρα και ειλικρίνεια έναντι της Λευκορωσίας, Μπελαρούς. Φυσικά έχουμε μια κατάσταση στη Λευκορωσία, Μπελαρούς, που αφενός έχουμε το θέμα των επαφών και της διατήρησης επαφών με τις αρχές και την κυβέρνηση. Είναι αναγκαίο να έχουμε τέτοιες επαφές, αλλά ταυτόχρονα τι βλέπουμε. Έχουμε και τις αντιδράσεις έναντι εκείνων που διαδηλώνουν τόπου κατά του καθεστώτος. Και σε αυτούς θέλουμε να τίνουμε χείρα βοήθειας και να βοηθήσουμε. Αυτό αναμένουν και εκείνοι από εμά. Πάντα κάτι τέτοιο γίνεται όταν αφορούν οι συζητήσεις και τα Δυτικά Βαλκάνια ή την Ανατολική γειτονία. Και έτσι εκφράζουμε τη θέση μας όσον αφορά και κάποιες αραβικές χώρες με αυτόν τον τρόπο. Αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά. Όμως, σε σχέση με την έκθεσή μας, δεν μπορούμε να συντάξουμε έκθεση υποτελεσίγραφο, ας το πω έτσι, της αντιπολίτευσης. Ίσως είναι καλύτερο να προσεγγίσουμε περισσότερο, να είμαστε πιο κοντά στην αντιπολίτευση, όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις όπου έχουμε μια τόσο ομή και σκληρή δικτατορία στο καθεστώς, στην κυβέρνηση. Είναι καλύτερο αυτό από το να αποφεύγουμε να έχουμε σχέσεις με την αντιπολίτευση. Όμως από την άλλη πλευρά στην έκθεση πιστεύω πρέπει να πιέσουμε να εντάσσονται τα θέματα εκείνα τα οποία θέλουμε να πετύχουμε και μπορούμε να πετύχουμε στην Μπελαρούς. Πρέπει να βρισκόμαστε στο πλευρό του πληθυσμού των πολιτών. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να καταστήσουμε σαφές προς την κυβέρνηση ότι οι δικές μας δραστηριότητες έναντι των αρχών θα είναι μια σκληρή στάση. Όταν υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι, πολιτικά όταν υπάρχουν διώξεις, ε, ομές διώξεις και ομή καταστολή και όταν τα πράγματα επιδεινώνονται και όταν τις σχέσεις μας με τις αρχές αυτές της Λευκορωσίας στην περίπτωση αυτή αν χαλαρώσουμε αυτή τα, αυτά τα σκληρά αιτήματα και τις διεκδικήσεις μας, τότε θα είναι ένα λάθος μήνυμα προς τους πολίτες. Να το επαναλάβω για άλλη μία φορά. Ευχαριστούμε όλοι τον εισηγητή για αυτή την έκθεση και μπορούμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, παρότι μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Αλλά η έκθεση θα πρέπει να πω και κάποιες τροπολποιήσεις πρέπει να ε, τύχουν στην έκθεση αυτή. Δηλαδή πιο σκληρή αντιμετώπιση των αρχών της Λευκορωσίας από πλευράς μας, από πλευράς των ετοιμάτων μας. Θέλω να το υπογραμμίσω αυτό έναντι των πολιτών των, της Μπελαρούς. Είμαστε υπέρ άμεσων επαφών και αυτό το μήνυμα πρέπει να είναι ένα σαφές μήνυμα έτσι όπως θα το αποστείλουμε. Είμαι πεισμένος ακράδαντα ότι με βάση αυτά που η συντάσσει και έχει εντάξει στην έκθεσή του. Αυτά πρέπει να εκφράσουμε και να τονίσουμε. Να τα επανεκπονήσουμε, να τα αναδιατυπώσουμε ώστε η θέση μας έναντι της Μπελαρούς να μπορεί να επιτευχθεί. Και κάτι άλλο επιπλέον. Δεν θέλουμε με κανένα τρόπο η αντιπολίτευση τις θέσεις της, ας το πω έτσι, να επηρεαστούν κάποια πράγματα. Όχι, η κατάσταση είναι τόσο έντονη και υπό τέτοια πίεση και τεταμένη στην Πελαρούς που πρέπει να έχουμε την ευαισθησία στις δράσεις μας και στις, στα διαβήματα που αναλαμβάνουμε και στις δραστηριότητες μας εκείνους να υποστηρίξουμε που πραγματικά βρίσκονται και σε αντιπαράθεση με το καθεστώς της Μπελαρούς. Κύριος Πέτερινγκ, παρακαλώ. Äh, äh, Σα ευχαριστώ. Είναι ωραίο να λαμβάνω τον λόγο μετά τον Γιέζι Μπούζεκ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παλέτσκι θερμά για την έκθεσή του αυτή. Και έχουμε νομίζω όχι μόνο πολιτική αλλά και ηθική υποχρέωση να βρεθούμε στο πλευρό των πολιτών της Λευκορωσίας. Και μια άλλη πτυχή να αναφέρω αν έχει ήδη προαναφερθεί, ζητώ να δείξετε κατανόηση. Αλλά θέλω να το υπογραμμίσω έστω για άλλη μια φορά. Στη Βίλνιους, την πρωτεύουσα της Λιθουανίας, υπάρχει το εξόριστο πανεπιστήμιο των ε, ε, ανθρωπιστικών επιστημών European Humanities University. εκεί σπουδάζουν και νέοι από τη Λευκορωσία παράκλησή μου ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωκοινοβούλιο να ενδιαφερθούμε για αυτούς τους φοιτητές ε, και να τους βοηθήσουμε και χρηματοδοτικά να τους υποστηρίξουμε. Είναι εξαιρετικοί οι άνθρωποι και είπαν όταν πάτε στο Βίνιους ε, μην ξεχάσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό αυτό το ακαδημαϊκό όργανο. Θέλουμε μια μέρα να ζούμε σε ένα ελεύθερο καθεστώς. Και κατά τούτο λοιπόν αν αυτό δεν έχει ήδη ληφθεί υπόψη να, να το τονίσουμε σε σχέση με την έκθεση του κυρίου Σε ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Σάιρος Βόλσκι παρακαλώ. <clears throat> Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Κάποιες φορές τα πολλά διπλωματικά λόγια καταλήγουν σε κενή διπλωματία. Θα είμαι λοιπόν ε, σαφής. Εγώ δεν είμαι ευγνώμων προς τον ε, εισηγητή. Είμαι μάλιστα πολύ αντίθετος με τα όσα λέει η σύσταση. Όπως είπε ο κύριος Παλέτσκι στο Ευρωκοινοβούλιο, έχει μιλήσει για τη Λευκορωσία 37 φορές τα τελευταία χρόνια και για πρώτη φορά η έκθεση στο πρώτο σχέδιο απέχει από τη σταθερή γραμμή και λαμβάνει απόσταση από τη σταθερή γραμμή του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν θα μιλήσω για τα τμήματα της έκθεσης με τα οποία συμφωνώ. Είναι σωστά και από ποσοτικής ε, πλευράς είναι η πλειοψηφία. Αλλά με ενδιαφέρουν αυτά τα οποία είναι αρνητικά για μένα. Όχι απλώ λοιπόν αποχωρεί από την σταθερή γραμμή του Κοινοβουλίου, την επιχρόνια σταθερή γραμμή μάλιστα, αλλά διαπράττει κάποια μαρτήματα για να μην τα πω παραπόματα, αντιφάσκει με τη σταθερή γραμμή του Κοινοβουλίου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είμαστε συνεπεί. Έπειτα, αντιφάσκει με την πραγματικότητα στην ε, Λευκορωσία. Για πρώτη φορά το Ευρωκοινοβούλιο και ο εισηγητή του παίρνει το μέρο των ε, επισήμων του Μίνσκ, λέγοντα ότι η βελτίωση τη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, είναι σημαντική, πράγμα που δεν εληθεύει. Και μάλιστα προτείνει την άρση των κυρώσεων που έχουν ε, επιβληθεί στη Λευκορωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα ομόφωνα. Οπότε δεν αμφισβητεί μόνο την πάγια γραμμή του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά στην πολιτική της. Ουσιαστικά αμφισβητεί το ίδιο το δόγμα της πολιτικής μας ε, με διπλά μέτρα και διπλά σταθμά. Κυρώσεις για δημοκρατικές συμπεριφορές σε κυβερνήσεις, αλλά άνοιγμα προς τους πολίτες, την κοινωνία. Η κατάσταση τη δημοκρατία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχει αλλάξει. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι υπάρχει αλλαγή. Όπου κι αν ε, κοιτάξει κανεί από την κατάρρευση τη δημοκρατική αντιπολίτευση και μετά. Είναι φυλακισμένοι οι άνθρωποι αυτοί. Το ίδιο και ο υποψήφιος για το βραβείο Ζαχάροφ ε, του σώματος εδώ. οι πολιτικοί κρατούμενοι είναι ακόμα στις φυλακές. Και σήμερα κιόλας υπάρχει διχασμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο σώμα μας και ούτως ή άλλως για μας η κόκκινη γραμμή ήταν πάντοτε η πολιτική κρατούμενοι. Η Παλάτα, το κοινοβούλιο τη χώρα δεν αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνον. Έχουμε πολλέ επιφυλάξει ω προ την ε, δημοκρατία και σε πολλά άλλα κράτη, αλλά για το συγκεκριμένο κράτο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν εκπροσωπείται καν στην Euronest. Πρόσφατα ήμουν στην ομάδα εργασία, χθε μόλι μάλλον ήμουν στην ομάδα εργασία για την Λευκορωσία τη Euronest. Και η θέση των περισσότερων είναι ότι οι βουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και των υπόλοιπων συμμετοχούσων χωρών έχουν ιδιαίτερα επικριτική στάση για τόσα συμβαίνουν στη Λευκορωσία. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που έξι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ηγέτες ε, των κομμάτων ηγέτε των οποίων βρίσκονται στη φυλακή. Θεωρούν την έκθεση αυτή σκανδαλώδη. Κύριε Ισηγητά, ε, επικαλεστήκατε την αρχή more for more, περισσότερα για πορό, περισσότερα. Αλλά εσεί προτείνετε το more for less, περισσότερα για λιγότερα. Καλό λοιπόν του ε, ευρωβουλευτέ από τα νέα κράτη-μέλη που ακόμα θυμούνται τον αγώνα του για τον εκδημοκρατισμό και την ελευθερία και περιμέναν στήριξη από την τότε Ευρωπαϊκή Ένωση, την τότε Ευρώπη, να, να θυμηθούν πόσο πολύ θέλανε την πολιτική μας στήριξη και πόσο εμείς όμως αισθανθήκαμε προδομένοι όταν δεν λάβαμε τη στήριξη αυτή. Ευχαριστούμε κύριε Βόλσκι. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω τώρα να κρυγορήσω. Τα πάνε περισσότεροι συνάδελφοι. Μια ερώτηση έχω προς τον εισηγητή. Σε σχέση με αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Αρής Βόλσκι. Λέει η έκθεση πως το 2012 είχαμε βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Παλέτσκης να το εξηγήσει αυτό. Γιατί πραγματικά απορώ να διαβάζω κάτι τέτοιο. Δεν θα μου κάνει εντύπωση παραδείγματος χάρη να μιλούσαμε για επιδείνωση της κατάστασης. Γι' αυτό θα ήθελα να μας πει ο κύριος Παλέτσκης τι εννοεί εδώ πέρα. Ότι το 2012 είχαμε βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν το καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ. Καλή ερώτηση. Ο κύριος Λαντσμπέργης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω κάποιε παρατηρήσεις. Μία για τις προθέσεις. και τον πολιτικό διάλογο. όπου μιλάμε για κύρωση της απαγόρευσης βίζας για σημαντικά, σημαντικούς αξιωματούχους της Λευκορωσίας και δηλαδή το να ακυρωθεί η απαγόρευση αυτή η βίζας είναι ήδη κάτι το κακό. Γιατί δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή, καμία βελτίωση, δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με την ατιμορρησία, αλλά εμείς προτείνουμε να σταματήσει αυτό και να διευρύνουμε και τις επαφές με τους αξιωματούχους. Τους αξιωματούχους. Τους αξιωματούχους που έχουν τιμωρηθεί με απαγόρευση εισόδου τώρα θα έχουμε περισσότερες επαφές. Υπάρχει κάποια αντίφαση και είναι και κατά των αρχών μας. Και βεβαίω ε, χάνουμε και το μοναδικό μέσο που έχουμε για να επηρεάσουμε τις εξελίξεις καλό θα ήταν να έχουμε και πιο ξεκάθαρη διατύπωση. Εκεί που μιλάμε για τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου. Μα δεν γίνονται εκλογές. Ε, οπότε καλό να μην χρησιμοποιούμε τέτοιες διατυπώσεις. Καλό είναι τι να παρακινήσουμε τις, εκλογές, να τις αρχές να γίνουν εκλογές αντί για ε, διορισμοί. Το ίδιο πρέπει να γίνει και για τη Ρωσία βεβαίως, αλλά τώρα με τη Λευκορωσία έχουμε περισσότερο θάρρος και πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οπότε το να μιλάμε για μεταρρυθμίσεις του εκλογικού νόμου όταν δεν υπάρχουν εκλογές ας είμαστε ειλικρινείς. για τις μειονότητες. Δεν υπάρχει κάποια σύσταση για ίσως όρους. Το, ε, το θέμα εδώ πέρα αφορά την επιβίωση. Μιλάτε για λιθουανική μειονότητα στις ε, περιοχές που συνορεύουν το θέμα δεν αφορά ε, ίσους όρους, αλλά την ίδια την επιβίωση. Ειδικά όταν υπάρχουν περιοχές όπου προγραμματίζεται ένας νέος, ένα νέο περνικό εργοστάσιο. Οπότε θα αλλάξει τελείως αυτή η περιοχή. Η δημογραφία της, η οικονομία της, Και ίσως, δεν ξέρω, ο στόχος είναι να φύγει αυτή η μειονότητα. Και πρέπει η Λευκορωσία να τηρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας στους πυρηνικούς σταθμούς. Δεν είναι γενικό, κύριε Λαντσμπέργκης, λέει ο πρόεδρος. Και, κοιτάξτε, μιλάμε για νέους πυρηνικούς σταθμούς 30 χιλιόμετρα από το Βίλνιους, από την πρωτεύουσά μας. Πρωτεύουσα ενός κράτους μέλους απαράδεκτο. Και θα έπρεπε να είναι απαράδεκτο και για την Ένωση. Δεν αναφέρεται έτσι πουθενά. Καμία κριτική. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λαντσμπεργκής, αλλά πρέπει να κλείσει η συζήτηση πολύ γρήγορα κύριε Νέιτς και μετά ο εισηγητής. Ε, ναι, δεν είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στην αντιπροσωπεία μου το σχέδιο σύστασης με ε, πολλές λεπτομέρειες, αλλά η ενεξελίξη συζήτηση δείχνει ότι η θέση του εισηγητού δεν ε, είναι κάτι που συμμερίζονται οι περισσότερες αντιπροσωπείες ή τέλος πάντων πολλά μέλη της Επιτροπής. Κοιτάζοντας το χρονοδιάγραμμα και βλέποντας ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η επόμενη εβδομάδα, 5 Ιουνίου, το μεσημέρι. Σκέφτομαι, δεν θα έπρεπε να παραταθεί αυτή η περίοδος να αναβληθεί η προθεσμία ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε και με άλλου συναντέλφους και αντιπροσωπείε. Διότι θα είναι σε πολύ άβολη θέση ο εισηγητή όταν ε, καταψηφιστεί η έκθεσή του ή εάν καταψηφιστεί γιατί η πλειοψηφία των υπόλοιπων μελών δεν την αποδέχεται. Από τη μια ε, συνάδελφη πρόεδρε καταλαβαίνω την ε, συγχυσή μας σε σχέση με τη Λευκορωσία και την ματέωση που αισθανόμαστε. Οι περισσότεροι έχουμε την αίσθηση ότι έχουν γίνει πολλές απόπειρες, πολλές προσπάθειες και τίποτα δεν έχει αποδώσει. Αυτό θα πρέπει να μας εμπνεύσει να πούμε να αλλάξουμε πορεία ενδεχομένως αλλά τώρα σε μια σύνοδο πριν την καλοκαιρινή διακοπή να ληφθεί τέτοια απόφαση, όχι, να αναβληθεί η προθεσμία, να δοθεί περισσότερος χρόνος για τις τροπολογίες και όσοι γιατί σας σκεφτεί να γίνει ψηφοφορία ούτε καν το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια, ίσως και αργότερα, ώστε να υπάρχει μια συνενετική προσέγγιση. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν θα ήταν καλό για το Κοινοβούλιο συνολικά να απορριφθεί το σχέδιο έκθεσης. Και νομίζω ότι ακούγοντας ε, όλες αυτές τις αντιδράσεις σήμερα, κάτι τέτοιο μπορούμε να φανταστούμε. Αυτό θέλω να πω. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για αυτή την ε, πρόταση. Όντως μπορούμε να αναβάλουμε ως τις 12 Ιουνίου την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Οι τροπολογίες αν γίνεται όμως να είναι στα αγγλικά. Κύριε Βόλσκι, είναι εδώ ο Υπουργό. Αν έχετε μόνο μια πρόταση να πείτε. Μια ε, κουβέντα. Ναι, ε, να αναβληθεί η τροπολογία και να περιμένουμε στον Οκτώβριο. Να προσκληθεί η Λευκορωσία στη Σύνοδο. Κύριε Παλέτσκη, ο εισηγητή, πολύ σύντομα, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, όπω προέβλεπα. Το θέμα αυτό είναι θερμό. Ε, είμαι ανοιχτό σε κάθε άποψη και ευχαριστώ όλους όσους τοποθετήθηκαν. Όμως... Το σημαντικότερο είναι ότι υπήρχε συμμετοχή στη συζήτηση. Να τονίσω εδώ και πάλι ότι είχαμε πάρα πολλά ψηφίσματα, έγγραφα για τη Λευκορωσία, τα οποία αντιδρούσαν στα α, δυσάρεστα γεγονότα που ελάμβαναν χώρα στη χώρα αυτή. Είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 9 χρόνια που εγώ είμαι μέλος του Κοινοβουλίου, που επιτέλους συζητούμε την κατάσταση στη Λευκορωσία. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτό θα είναι ένα μεγάλο ε, συν για το Κοινοβούλιο. Και ως προς κάποιες ερμηνείες που ακούστηκαν, νομίζω οι συνάδελφοι δεν είχαν αρκετό χρόνο για να διαβάσουν την έκθεση. Διότι υπήρχαν, ακούστηκαν δηλώσεις που δεν αντικατοπτρίζουν καθόλου το περιεχόμενο της έκθεσης. Ως προς την ερώτησή σας, να επαναλάβω αυτά που είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση. Γιατί χρησιμοποιήθηκε αυτή η διατύπωση. Μπορώ να σας το εξηγήσω πάντως και κατηδίαν. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό να αναβληθεί. Να παραταθεί η περίοδος για την υποβολή τροπολογιών. Από την άλλη, ταυτόχρονα καλό θα ήταν η θέση του Κοινοβουλίου να έχει παγιωθεί πριν την Σύνοδο του Βίλνιους. Εάν γίνεται λοιπόν να συμβαδίσουμε και με, το, να, με αυτό το γεγονός θα ήταν καλό. Ξέρω ότι χρόνος δεν υπάρχει και γι' αυτό ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή τους. Ευχαριστώ ιδιαίτερος τους Κιώδης και μάλιστα τον κύριο Προτασέβιτς με τον οποίο έχουμε διαρκώς ε, επικοινωνία. Συζητήσαμε κάποιες από τις θέσεις μας και πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Να διορθώσουμε τα σημεία που δεν αρέσουν σε όλους και η έκθεση αυτή να αντικατοπρίζει πραγματικά την γραμμή του Κοινοβουλίου. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα είναι εφικτό, πιστεύω. Ευχαριστώ κύριε Παλέτσικη, Πρώτα απ' όλα αποφασίσαμε παράταση της περίοδου για την υποβολή τροπολογιών μέχρι τις 12 Ιουνίου το μεσημέρι. Και μετά θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το χρονοδιάγραμμα. Και τώρα κλείνουμε με το σημείο αυτό. Περνάμε στο επόμενο. Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων του Μπαγκλαντέ. Σύντομη παύση.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 Ε, μπορεί να είστε λίγο κουρασμένοι, αλλά έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Τη συζήτησή μας με την Υπουργό Εξωτερικών του Μπαγκλαντές. Την κυρία Ντίπου Μόνη για τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα. Σας καλωσορίζω. Είστε και η πρώτη γυναίκα υπουργό εξωτερικών τη χώρα σα. Είστε ταυτόχρονα μία από τις δύο γενικούς γραμματείς του κόμματος Αβάμι League κατά το οποίο δείχνει πως ε, επηρεάζεται τα όσα συμβαίνουν στη χώρα σας. Σαφώς. πολύ περισσότερο πώ μπορεί η Υπουργό Εξωτερικών. Εκτιμούμε βεβαίω αυτά τα οποία έχετε κάνει για τα δικαιώματα των γυναικών, την πολιτική της υγείας και τις κοινωνικές εξελίξεις και την κοινωνική εξέλιξη και βεβαίω μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας πώς έχει η κατάσταση στον τομέα της ε, με την υπόθεση του κτηρίου που κατέρευσε με τις κοινωνικά ζητήματα, δικαιώματα των εργαζομένων, εμπορική πολιτική, αναπτυξιακές δυνατότητες και το πώς θα συνδέσουμε τον Παγκλαντές με τις σχέσεις μας και βεβαίω μας ενδιαφέρουν και οι εξελίξεις στη χώρα σας αν με ενημερώνουν σωστά θα έχετε εκλογές φέτος. Γι' αυτό χαίρομαι για το ότι έχουμε την ευκαιρία να έχουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ξεχωράτε, Κύριε Μπροκ, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας την ιδιαίτερη εκτίμησή μου για την ευκαιρία που μου δίνετε να συνομιλήσω με την Επιτροπή σας. Ε, κάποιοι από εσά έχουν έρθει στο Μαγκλαντές και περισσότεροι έχετε κάποια σχέση με τα θέματα του Μαγκλαντές. Στην Δύση γενικότερα και στην Ευρώπη το Μπαγκλαντές ε, δεν ε, υπάρχει στην δημόσια συζήτηση ως κάτι το θετικό. Για να είμαι ειλικρινής, καμιά φορά όταν εμφανίζεται το Μπαγκλαντές στις ειδήσει είναι μόνο για καταστροφές ή κάτι παρόμοιο, αλλά υπάρχει βεβαίως, υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα που συμβαίνουν στο Μπαγκλαντές. Μπορεί πολλοί από εσά να γνωρίζετε κάποια από αυτά τα πράγματα και να έχετε επαφή με τους πανεπιστημιακούς και την κοινωνία των πολιτών, θα ήθελα παρόλα αυτά να αναφέρω κάποιες πτυχές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Πριν από 42 χρόνια, όταν γεννήθηκε το Μπαγκλαντές ε, από έναν πόλεμο, πάρα πολλοί ήταν επιφυλακτικοί για την επιβίωση του νέου εθνικού κράτους και θεωρούσαν πως με τεράστιο πληθυσμό και σχεδόν καθόλου πόρους το, στο Μπαγκλαντές θα έδινε αγώνα. Χάρη λοιπόν στην επιμονή του λαού μας ε, καταφέραμε να επιτύχουμε και να διαψεύσουμε ε, τους επικριτές μας και προοδεύσαμε σε όλους τους τομείς. Την τελευταία δεκαετία η οικονομία μας ε, είχε αύξηση του ΑΕΠ κατά 6% κατά μέσο όρο, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος είχε κρίση. Θεωρούμε τώρα πως είμαστε μια οικονομία με πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης. Πάρα πολύ Επίσης ε, σημαντικά ήταν τα κοινωνικά επιτεύγματα. Επιτύχαμε κάποιους στόχους της χιλιετίας ε, σχεδόν 6 με 7 χρόνια πριν από την πρωτισμία. Δεν θέλω να μπω τώρα στα στοιχεία, απλά να σου πω πως αυτά φαίνονται στον αριθμό του παιδιών που πάνε σχολείο, το μείωση του αριθμού των παιδιών που πέφτουν, μείωση της παιδική νησιμότητας, της βρεφικής νησιμότητας και της νησιμότητας των γυναικών στην Ε, Βλέπουμε πως ο αλφαβητισμό περιορίζεται στο 1 τέταρτο του πληθυσμού, όλα τα κορίτσια γράφονται στο σχολείο και συχνά πάνε καλύτερα από τα αγόρια. Οπότε βλέπουμε καλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία, σε αστικές αλλά και μη αστικές περιοχές, καθώ επίσης και στον τομέα της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Πριν από λίγα χρόνια δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τέτοια πράγματα στον Μπαγκλαντές. ξεχωρίζει το Μαγκλαντές γιατί έχουμε επιτύχει τόσο σημαντική κοινωνική πρόοδο ακόμα και με χαμηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό αναγνωρίζουν πάρα πολλοί ερευνητές. Βεβαίως ε, συνεχίζουμε να ζητάμε αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά νομίζω πως θα μπορούσαμε να επιτύχουμε πολύ περισσότερα με τις τοπικές ιδέες, τους δικούς μας πόρους στην εκπαίδευση και την εκπαίδευση στα θεσμικά μας όργανα. Θα ήθελα να φέρω άλλο ένα παράδειγμα, παραδείγματος χάρη τη διαχείριση των καταστροφών. Κάτι το οποίο φάνηκε αυτό τον μήνα, καθώς αντιμετωπίσαμε έναν τροπικό κυκλώνα με μόλις 38 νεκρούς. Έχουμε τεράστιο πληθυσμό, πάρα πολύ νέο, πειθαρχημένο, εργατικό και αυτό αναγνωρίζεται και για τα 6,5 εκατομμύρια μετανάστες που υπάρχουν από ολόκληρο τον κόσμο, αλλά βεβαίως και από την εργατικότητα του λαού μας. Αυτά τα λέω μόνο ως παράδειγμα, βεβαίως οι πανεπιστημιακοί έχουν να πούν πολλά περισσότερα. Αυτό το οποίο μας ενώνει με την ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολλά πράγματα. Στην πορεία της χώρας μας από το 1972 λάβαμε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρσι σημαδεύσαμε τα 40 χρόνια συνεργασίας ε, και οι σχέσεις μας εμβαθύνονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος ε, χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας στο Μπαγκλαντές, ε, μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και μεγαλύτερος εισαγωγέας προϊόντων του Μπαγκλαντές. Είχαμε λοιπόν και μία συμφωνία πλαίσιο για τη συνεργασία μας που κάλυπτε εμπορικές σχέσεις, ανθρώπινα δικαιώματα, περιβαλλοντικά ζητήματα και ασφάλεια διατροφική. Μετά την τελευταία διαβούλευση το Δεκέμβριο του 2012 στις Βρυξέλλες πλησιάζουμε στο να έχουμε μία πολιτική διαβούλευση. Σαφώς λοιπόν οι σχέσεις μας βασίζονται σε αξίες όπως η ειρήνη, η ελευθερία, το κράτος δικαίου, η ανοχή, η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό επιτρέπει στον Μπαγκλαντές και την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργάζονται από τον ΟΗΕ μέχρι τον ΑΣΕΜ για ζητήματα όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, κλιματική αλλαγή και αντιτρομοκρατία. Όπως είπα τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερο εισαγωγέα προϊόντων μας. 56% των εξαγωγών μας πάνε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα εξάγουμε από ε, ρούχα μέχρι πλοία. Επίσης κατεψυγμένα δερμάτινα προϊόντα, ε, ελαφρά βιομηχανικά προϊόντα όπως ποδήλατα, αλλά και λογισμικό. Τα προϊόντα μας έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τις σχετικές συμφωνίες. Βεβαίω βασικό τομέα είναι η κλωστοϊφαντουργία που απασχολούνται 4 εκατομμύρια άτομα και 20 εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από αυτήν. Αν σκεφτούμε και τις σχετικές με τις μηχανίες, όπως τις βαφές, τη συσκευασία κτλ. Μιλάμε για ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά τα τελευταία δέκα χρόνια, η βιομηχανία αυτή έχει συνεισφέρει σε σημαντικές κοινωνικές αλλαγές στην χώρα. Βοήθησε να απελευθερώσει γυναίκες από πολύ φτωχά νοικοκυριά, από μια οικονομία χωρίς χρήμα ή τον παραδοσιακό ρόλο της νοικοκυράς. Πρόκειται για πράγματα λοιπόν τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούν και έχουν αλλάξει οι ρόλοι. Δηλαδή μετασχηματίζεται η παραδοσιακή, ο παραδοσιακός ρόλος γυναίκας ο οποίος ήταν αυτός της μη προσωπικότητας. Τώρα γνωρίζουν οι γυναίκες ότι έχουν δικαιώματα και μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις. Κυρίες και κύριοι, με βάση όλα αυτά τα οποία σας είπα, ε, τελευταία έχει αποτελέσει η βιομηχανία, η κλωστοϊφαντουργική του σε ένα αντικείμενο που απασχολεί την Ευρώπη μετά τα τελευταία ατυχήματα. Μετά από τα ατυχήματα αυτά, εμείς ε, προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε ε, τα ζητήματα τα οποία αφορούν αυτόν τον τομέα. Και πριν από αυτή την τραγωδία είχαμε σχηματίσει μια δεκαμελή επιτροπή πρώτη φορά στην χώρα κλαδική για να υπάρχει ασφάλεια στον χώρο εργασίας, πυρασφάλεια και τα λοιπά. Επίσης τροποποιήθηκε η εργασιακή νομοθεσία η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από την τραγωδία αυτή, Γιατί υπήρχε ξαφνική ανάπτυξη αυτού του κλάδου, κάτι το οποίο οδήγησε σε, κάποιες, σε κάποια εργοστάσια τα οποία δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές. Αυτό πρέπει να διορθωθεί. Εδώ πέρα η κυβέρνησή μας συμφωνεί με τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί κάθε ζωή είναι πολύτιμη. Μετά το ατυχημα στο Σαβάρ, αναλάβαμε κάποιες ε, μέσο και βράχοι πρόθεσμες πρωτοβουλίες. Υιοθετήθηκε μια τρικοματική ε, διακήρυξη, αλλά και διακήρυξη από κοινού με τους ε, εργαζόμενους και τους εργοδότες. Εργαζόμαστε λοιπόν για να προσληφθούν ακόμα 200 επιθεωρητές ε, εργασίας ε, και υπάρχουν τα σχετικά κονδύλια και η σχετική νομοθεσία θα πέρασε από το Κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Ο νέος νόμος θα επιτρέψει στους εργαζόμενους το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε ε, του συνέρχεστε σε λογικές διαπραγματεύσεις και για το ζήτημα των μισθών έχει σχηματιστεί επίσης μια σχετική επιτροπή. Για πρώτη φορά η Κλαδική Ένωση των Βιομηχάνων ζήτησε από όλα τα μέλη της να υποβάλουν εκθέσεις ε, επιθεωρητών, ε, επαγγελματιών επιθεωρητών για διάφορες ε, βιομηχανικές ζώνες και όσα εργοστάσια δεν κρυθούν κατάλληλα θα μετακομίσουν. Βεβαίως όλα αυτά κοστίζουν. Υπολογίζουν διάφορες οργανώσεις ε, πως για να συμμορφωθούν όλα τα εργοστάσια απαιτούνται 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ μεγάλο αυτό το νούμερο. Εάν σκεφτούμε ότι μπορεί να διατεθεί σε 5 χρόνια, σημαίνει πως ε, αντιστοιχεί σε 10 cents παραπάνω κόστος για το κάθε ρούχο που βγαίνει από εκεί. Νομίζω πως οι καταναλωτές στη Δύση μπορούν να το πληρώσουν αυτό ή και λίγο παραπάνω για τα εκατομμύρια γυναίκες που ράβουν για αυτούς σε μια μακρινή χώρα. Γι' αυτό καλωσορίζουμε τις ε, δεσμεύσεις ε, της Ένωσης Εργαζομένων στον τομέα αυτών για να τηρηθεί αυτή η συμφωνία. Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους τους εργαζόμενους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει ήδη τη στήριξή της και θα ζητούσα από το Κοινοβούλιο να μας στηρίξει σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία. Ίσως αν είχε γίνει αυτή η συζήτηση νωρίτερα, ε, όλοι θα είχαμε κάνει πολύ περισσότερα. Κυρίε και κύριοι, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, επίσης, που επηρεάζει αρνητικά τον Μπαγκλαντές σε μέρος του ε, ευρωπαϊκού τύπου και αφορά τα εγκλήματα πολέμου. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για το Μαγκλαντές είναι ένα μαγκλαντεσιανό δικαστήριο και σκοπεύει να δικάσει τους δράστες μιας ε, φρικτής γενοκτονίας και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας του 20ου αιώνα που διαπράκτηκε το 1974. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας ε, στην απόφαση, την πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου, η οποία ξεκαθαρίζει πως δεν υπήρχε ε, πολιτικό κίνητρο για αυτές τις ε, δίκες, όπως έλεγαν κάποια μήμιε. Ο εισαγγελέας κατέδειξε πως κανένας κατηγορούμενος δεν κατηγορήθηκε ε, για πολιτική δραστηριότητα παρά μόνο για τα φρικτά εγκλήματα που διέπραξαν κατά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Πράγματι υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο ε, για τις δίκες αυτές. 40 ε, χρόνια μετά την ανεξαρτησία το Μπαγκλαντές δείχνει πως θέλει να τελειώσει η κουλτούρα της ατιμορρησίας αυτό είναι αυτό το οποίο εγώ περιγράφω ως η φρίκη της ατιμορρησίας. Μετά από 40 χρόνια, εκατομμύρια άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους και περίμεναν να αποδοθεί δικαιοσύνη, βρήκαν κάποια παρηγοριά. Το δικαστήριο με την απόφασή του επαναβεβαίωσε πως κανένα άτομο υπεύθυνο για αυτά τα εγκλήματα δεν μπορεί να συνεχίσει να ξεφεύγει από την ε, δικαιοσύνη και να συνεχίσει να υπάρχει η ατιμορρησία. Καθώς, όπως λέει, έτσι οι παλιές πληγές ε, εξακολουθούν να υποτροπιάζουν. Γι' αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω πως η διαδικασία αυτών των δικών εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτή και στη διάθεση του καθενός για να παρατηρηθεί. Φαντάζεται κανείς στην Ευρώπη πως θα ήταν η μεταπολεμική Ευρώπη χωρίς δίκες για εγκλήματα πολέμου. Θα μπορούσαν όσοι έκαναν αυτά τα εγκλήματα να κυκλοφορούν ελεύθεροι μαζί με τα θύματα και τις οικογένειές τους ή να έχουν και καρτικά αξιώματα. Σας διαβεβαιώ πως η διαδικασία είναι τελείως διάφανη και σωστή και τη τις ε, διεθνείς προδιαγραφές. Τίθενται έτσι ερωτήματα για το ότι είναι πιθανή η θανατική ποινή. Εξηγήσαμε πως η νομοθεσία μας το προβλέπει όπως και σε άλλα μέρη της Ασίας και αλλού. Καθώς αυτό προκύπτει από το ε, νομικό μας πολιτισμό και τις απαιτήσει της κοινωνίας και ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αντιληφθεί τη φιλοδοξία του λαού μας για δικαιοσύνη και να δεχτεί αυτή την διαδικασία λογοδοσίας. Κυρίες και κύριοι, το Μπαγκλαντέ ιδρύθηκε αν δει κανείς ε, το πώς ε, είχαμε ξεκινήσει όταν έγινε ανεξάρτητη η Ινδική Υποήπειρος με βάση τον πλουραλισμό και τη δημοκρατία. Αλλά προσφάτως από όταν ξεκίνησε η δίκη για τα εγκλήματα πολέμου είχαμε ανεπανάληπτη βία από πλευράς της ε, Τζαμάτ Αλ-Ισλάμι και της φοιτητική της παράταξης, κατά το οποίο ο λαός απέρριψε. Από όταν βγήκε η πρώτη απόφαση του δικαστηρίου, η ελάχιστη αυτή μειοψηφία ξεκίνησε μια επίθεση σε ολόκληρο το μήκος και το πλάτος της χώρας. Επιτέθηκαν σε ηλεκτρικά εργοστάσια, ναούς, α, μειονότητες θρησκευτικέ, ακόμα και κατά των δυνάμεων της τάξης δημιουργήθηκε χάος και σήμερα υπάρχει σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και την τάξη του Μπαγκλαντές και την εσωτερική ασφάλεια θα έλεγα. Παρά τις προκλήσεις η... Ε, τα σώματα ασφαλείας απάντησαν με πάρα πολύ μεγάλη υπομονή. Είναι σαφές πως ο στόχος είναι ένας, να υπονομευτεί η διαδικασία, η δίκη για τα εγκλήματα πολέμου και κάποιος θα χαρακτήριζε αυτές τις πράξεις ως τρομοκρατικές. Ενώ λοιπόν προσπαθούμε να περιορίσουμε την Τζαμάτ Αλισλάμι, τέλος Μαρτίου είδαμε μια ξαφνική ε, άνοδο του Χεφαζάτ Αλισλάμ που θεωρούν πως ε, προστατεύουν το Ισλάμ Ζήτησαν λοιπόν την δυνατότητα να συγκεντρωθούν σε κάποιους μεντρεσέδες, άδεια η οποία τους δόθηκε, αλλά μετά προσπάθησαν να καταλάβουν την ντάκα. Και χάρη στα ΜΜΕ όλος ο κόσμος μπορούσε να δει το πραγματικό τους πρόσωπο και τα 13 αιτήματά τους. Κατέληξαν σε τυφλή βία, καταστροφή δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας και έκαψαν ακόμα και το Ιερό Κοράνιο. Τελικά αυτό κατέληξαν σε τελείως βίες ε, πράξεις. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να τους απομακρύνει και να τους διαλύσει εκτός της Ντάκας, από όπου και ήρθαν άλλωστε. Έκτοτε ε, υπάρχει προπαγάνδα στα ε, κοινωνικά μέσα όσον αφορά τις τυχόν απώλειες. Οι απώλειες ήταν 11 άτομα μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός. Τη στιγμή που ετοιμάζεται να απογειωθεί το Μαγκλαντές οικονομικά, βλέπουμε να ε, εμφανίζονται κάποιες δυνάμεις που αμφισβητούν τα ε, βασικά θεμέλια της χώρας μας. Ε, τη στιγμή ακριβώς που αρχίζει και η ευρωπαϊκή βιομηχανία να αναγνωρίζει το Μπαγκλαντές, κάτι το οποίο φαίνεται και από ευρωπαϊκές εμπορικές αντιπροσωπείες. Οπότε οι εξελιξει αυτή ήταν ιδιαίτερως ατυχείς. Μπορούμε να δούμε τα αιτήματα της Χεφαζάτ και θα καταλήξετε πως στόχο έχουν να εκμηδενήσουν την κοινωνική πρόοδο που έχει επιτευχθεί και εσείς έχετε επενέσει. Είναι προσβολή προς την κοσμική ταυτότητα του Μπαγκλαντές και είναι τελείως αντίθετα τα αιτήματα με το Σύνταγμά μας και με τις αξίες μας και τις φιλοδοξίες και τα όνειρα του λαού μας και τις αρχές με τις οποίες ιδρύθηκε το Μπαγκλαντές το 1971. Το Μπαγκλαντές λοιπόν αντιμετωπίζει καιρούς δύσκολους και εδώ πέρα ακριβώς χρειάζεται τους φίλους του ε, στο πλευρό των 150 εκατομμυρίων κατοίκων του. Θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στις ε, επόμενες εκλογές. Όλοι γνωρίζετε τις εξελίξεις, ε, τη συζήτηση που υπάρχει, τη 15η τροποποίηση του συντάγματος. Να σας πω πως εμείς ε, ήμασταν πάντα υπέρ του διαλόγου. Τα έχει πει πολλές φορές, ο Πρωθυπουργός επανειλημμένα έχει προσκαλέσει την αντιπολίτευση σε διάλογο για να δούμε πώς θα μπορέσουν να διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Επίσης, η Πρωθυπουργό ζήτησε από την αντιπολίτευση να επανέλθει στο Κοινοβούλιο και να συζητήσουμε όλα τα θέματα εκεί. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να σκεφτούμε τα αιτήματα εντός των ορίων του συντάγματος και με βάση κάποια κοινή συνεννόηση. Η Πρωθυπουργό χωρίς καμία προϋπόθεση πήγε ακόμη παραπέρα και παρουσίασε ε, ε, το προσχέδιο για το πώς η κυβέρνηση θα μπορέσει να βοηθήσει την εκλογική επιτροπή στην ε, τρίμηνη προεκλογική περίοδο. Η υπηρεσιακή κυβέρνηση θα αποτελείται από προσώπους όλων των μεγάλων κομμάτων για να διασφαλιστεί πως θα είναι πραγματικά μερόληπτη. Υπήρχε αρκετά μεγάλη σύγχυση για το ζήτημα της υπηρεσιακής κυβέρνησης και της κατάργησης της με την 15η αλλαγή του συντάγματος. Αυτά με βάση μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ακολούθησε συζήτηση στην Επιτροπή τη σχετική του Κοινοβουλίου και αντιλαμβάνεστε βέβαια πως πρέπει να συμμορφωθούμε με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η διεξαγωγή των εθνικών εκλογών βεβαίως είναι, είναι ζήτημα της εκλογικής επιτροπής. Αυτό είναι πεποίθησή μα για να ενισχύσουμε ε, τις εκλογικές διαδικασίες ε, όπως σε κάθε άλλη δημοκρατία. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έχει διεξάγει επιτυχώς 5.636 ε, εκλογικές διαδικασίες, ε, δημοτικών εκλογών δηλαδή, και ούτε μία φορά δεν υπήρχαν καταγγελίες κακοδιαχείρισης, μεταξύ των οποίων και κάποιες εκλογές για αναπλήρωση εδρών στο Κοινοβουλίο το καταστατικό τη ορίζει πως η εκλογική επιτροπή είναι πλήρως ανεξάρτητη και μην ξεχνάμε πως ε, συστάθηκε μετά από τα διαβούλευση με όλα τα πολιτικά κόμματα. Γι' αυτό είμαστε νομίζω σε θέση οι επόμενες εκλογές να γίνουν με τρόπο δίκαιο και ελεύθερο με τη στήριξη της υπηρεσιακής κυβέρνησης που θα αποτελείται από ερετούς εκπροσώπους του λαού. Σίγουρα αντιλαμβάνεστε πως ε, έχει φτάσει η στιγμή να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα στις εθνικές εκλογές ε, οι οποίες, ε, τις οποίες θα διαχειρίζονται ερετοί εκπρόσωποι. Όπως είπα, γνωρίζω πως η διεθνής κοινότητα θέλει οι εκλογές να είναι μη βίαιες και χωρίς αντιπαραθέσεις. Θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους φίλους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη διεθνή κοινότητα πως το Μπαγκλαντές παραμένει ανοιχτό για οποιαδήποτε στήριξη στην εκλογική διαδικασία. Και άρα είμαστε ήδη σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δεχτούμε ανεξάρτητους διεθνείς παρατηρητές για να παρατηρήσουν αυτή τη διαδικασία πριν τις εκλογές, κατά τη διάρκεια των εκλογών και προφανώς μετά τις εκλογές. Κυρίες και κύριοι, καταλήγοντας ως μια νεαρή δημοκρατία και μια ανερχόμενη οικονομία, το Μαγκλαντές έχει και κάποιους περιορισμούς και προκλήσεις. Τονίζουμε όμως πως όλα αυτά είναι φυσιολογικά για οποιαδήποτε νεαρή δημοκρατία. Αυτό μας το διδάσκει η ιστορία παντού στον κόσμο και ελπίζουμε τελικά πως θα καταφέρουμε να επιτύχουμε αυτά τα οποία απαιτούνται. Αυτό το οποίο ζητάμε από εσά είναι στήριξη και ε, το να αντιληφθείτε την κατάσταση και εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. We have now first the vice chair of the Ο αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής ε, Ασίας. Ο κύριος Μιχάηλο, παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Is that okay? Or... Εντάξει κύριε Βάιλο. Κύριε Σταρμοντάρτο, ο κύριος Αταμούνταλτο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, πώς σωστά αναφέρατε, το Μπαγκλαντές ήταν στον τύπο ως πηχιαία είδηση, δυστυχώς για τους λάθος λόγους. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή, μια και από τη μία πλευρά έχουμε την τεράστια κλωστοϊφαντουργία στη χώρα σας, δεύτερη μετά από την Κίνα παγκόσμια. Και είναι μία από τις κύριες εξαγωγικές δραστηριότητες της χώρας σας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κλωστοϊφαντουργικά. Πιστεύω ότι 70% συνολικά πάνε στην Γερμανία από αυτά τα προϊόντα, δεν κάνω λάθος. Και εμείς όπως μπορείτε να φανταστείτε ανησυχούμε για αυτή την κατάσταση εκεί, διότι κατά κάποιο τρόπο είμαστε συνένοχοι στα όσα συνέβησαν κατά τις δύο αυτές καταστροφές που είχαμε στις ειδήσει τη φωτιά, την πυρκαγιά αφενός και τη δεύτερη φορά την κατάρρευση των κτηρίων. Και εμείς εμπλεκόμαστε διότι φυσικά υπό εμπορικούς όρους προσπαθούμε με κάθε τρόπο να έχουμε τις καλύτερες πιο προσιτές τιμές για τα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα, μειώνοντας έτσι το κέρδος, περιθώριο κέρδους για τους ε, επιχειρηματίες. Αλλά δυστυχώς από την άλλη πλευρά πρέπει να επισημάνουμε κάτι. Και αυτό είναι ότι παρότι έχουμε την καταστροφή σε σχέση με την πυρκαγιά, μια άλλη καταστροφή συνέβη και όπως επισημάνατε στη συνέντευξη τύπου που δώσατε στο κανάλι CNN, η κυβέρνησή σας κάνει ότι περνάει από το χέρι της για να προσπαθήσει και να αντιμετωπίσει αυτά τα οποία προηγούμενα έπρεπε να ρυθμιστούν και να αντιμετωπιστούν. Αν δεν κάνω λάθος, δεν ήταν πολύ εκείνοι οι επιθεωρητές. Ήταν έξι όλοι και όλοι, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να ήταν πολύ, μπορούσαν να ήταν περισσότεροι, αλλά νομίζω ότι σωστά κατευθύνεστε στην ε, ορθή κατεύθυνση ζητώντα να αναλυφθεί η δράση. Ένα άλλο θέμα στο οποίο αναφέρατε στο CNN είναι το θέμα των ελάχιστων μισθών και το θέμα του ελάχιστου μισθού είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση και ολοκληρώνω με αυτό ότι αυξάνοντας τον ελάχιστο μισθό θα έδινε την δυνατότητα σε εκείνους τους ανθρώπους που έχουν επενδύσει στην κλωστοϊφαντουργική ε, βιομηχανία παραγωγής ενδυμάτων να κάνουν αυτό το οποίο είναι σημαντικό για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε αυτόν τον κλάδο. Σας ευχαριστώ. Επικεντρώθηκα σε ένα μόνο θέμα επειδή πιέζει ο χρόνος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκάλερ, σας ευχαριστώ πολύ και καλώς ορίσατε Υπουργέ. Εδώ είμαι, δεξιά, στη δεξιά πλευρά. Καλώς ήρθατε κυρία Υπουργέ στην δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλωσορίζω όταν αναφέρατε τα θέματα των επιτευγμάτων όσον αφορά την πτυχή αυτή είναι ένα πολύ θετικό γεγονός και είμαι ικανοποιημένος στο ότι ρητά αναφερθήκατε στην κοσμική, στις κοσμικές τάσεις της ε, εγκαθίδρυσης ε, της χώρας σας, ε, του Μπαγκλαντές, είναι κάτι το οποίο συνδέεται με την διεξαγωγή και ελεύθερων και δημοκρατικών εκλογών και αυτό είναι κάτι που καλωσορίζουμε και υποστηρίζουμε απόλυτα στο Ευρωκοινοβούλιο εδώ. Αλλά από την άλλη πλευρά όσον αφορά την κοσμική μορφή του κράτους όταν η κοσμική εξουσία δεν είναι αποτελεσματική στρέφονται αλλού οι πολίτες και σε σχέση με το Πακιστάν όπου ένα θυγατρικό κόμμα, ένα αδελφό κόμμα το Αγουάμι διελήθη, κατέρευσε, βρισκόταν στην κοσμική συμπολίτευση και παρόλα αυτά διαλύθηκε. Δεν ήταν τα ριζοσπαστικά κόμματα εκείνα τα οποία πήραν το πάνω χέρι στο Πακιστάν, αλλά δείχνει την τάση και την μετάθεση, μετακίνηση ψηφοφόρων. Όταν οι οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για μεγάλα τμήματα του πληθυσμού είναι αρνητικές και όπως είναι και η κυβέρνηση δεν κάνει αυτό το οποίο πρέπει, όπως βλέπουν τα πράγματα οι ψηφοφόροι, τότε ριζοσπαστοποιούνται. Και αυτό είναι γεγονός παγκόσμια σε όλες τις χώρες. Γι' αυτό θα απίφθηνα έκκληση και σε σχέση τώρα με θέματα τα οποία αφορούν την κλωστοϊφαντουργία, όλα τα μέτρα τα οποία αναλαμβάνεται, να είναι πραγματικά αποτελεσματικά και να είναι συντονισμένα. Να ε, έχουμε με βάση το νόμο συμφωνίες και όρους που θα εφαρμόζονται και ο νόμος θα εφαρμόζεται. Ερώτηση. Σε σχέση με τις προδιαγραφές ε, του ε, Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας είσαστε πλήρες ε, μέλος και έχετε προσυπογράψει αυτές τις, ε, ε, αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και θα υπάρχει το δικαίωμα και πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα διοργάνωσης σε συνδικάτα των εργαζομένων και ελεύθερης δράσης των συνδικάτων και ελάχιστων μισθών που θα συναποτελούν μέρος του συνολικής συμφωνίας, του συνολικότερου πλαισίου. Αυτό όμως που εμείς μπορούμε να κάνουμε εδώ είναι να ασκήσουμε πίεση στις δικές μας ευρωπαϊκές εταιρείες. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη, υπευθύνη υπευθυνότητα από πλευρά μα. Ε, όχι μόνο να προσπαθούν να πετύχουν τι χαμηλότερε εφικτέ τιμέ, αλλά να συνειδητοποιήσουν ε, οι πολίτε μα ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Δεν μπορούμε μόνο να πληρώνουμε τι χαμηλότερε τιμέ ε, για τα ενδύματα και τα κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα. Είναι λοιπόν και η δική μα δουλειά που πρέπει εμεί να κάνουμε, αλλά και εσεί το δικό σα μέρο τη δουλειά για του πολίτε σα. Ευχαριστώ. Κυρία Κυρία Ντεκεζέρ, ευχαριστώ πρόεδρε. Η κυρία Ντεκεζέρ, ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ. Πράγματι, θεωρούμε τη χώρα σας ως μια χώρα που μας είναι ιδιαίτερα συμπαθής και της δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή. Το ψήφισμα για τον Μπαγκλαντές που ψηφίστηκε στην ε, περασμένη Ολομέλεια του Στρασβούργου απασχόλησε πολύ τις συζητήσεις των βουλευτών και έδειξαν αυτοί ότι έχουν ε, συνείδηση ότι το επεισόδιο το πρόσφατο με την κατάρρευση του κτηρίου ήταν κάτι που αφορά ευθύνη πολλών διαφορετικών ε, μερών. Βεβαίω οι αρχέ του Μπαγκλαντέ έχουν ευθύνη, αλλά και εμεί ω καταναλωτέ και η Ευρώπη, τη οποία δραστηριοποιούνται εταιρείε εκεί, έχουμε ευθύνη. Κοίταξα και εξέτασα με προσοχή τα μέτρα που λάβατε και θέλω να σας πω ότι και σε εμά στην Ευρώπη από την αρχή της ευρωπαϊκής διαδικασίας η πρόοδος σε θέματα νομοθεσίας που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία και σε εμά η αφορμή συνήθως ήταν μεγάλα ατυχήματα, κυρίως σε ορυχεία. Ε, έτσι συνειδητοποίησαμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Είμαι λοιπόν και εγώ βέβαιη ότι θα προοδεύσετε με τη σειρά σα και στη δική σα χώρα. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Στην νομοθεσία σα έχετε κάτι που να αφορά την αλυσίδα υπεργολαβιών συνεργατών δηλαδή, γιατί αυτό έχει σχέση με τα όσα συνέβησαν, με το πρόσφατο δράμα. Υπήρχε μια μυριάδα υπεργολάβων και ήταν δύσκολο να εντοπιστεί και να λογοδοτήσει ο πραγματικά υπεύθυνο. Και έπειτα, για όσους δεν ε, αποδέχτηκαν την συμφωνία που συνήθι το Μάιο, τι θα κάνει η κυβέρνηση ως προς εκείνους. Και τέλος, είστε μια χώρα νεαρή η νομοθεσία σα για θέματα υγιεινής και ασφάλεια στην εργασία πόσο έχει προχωρήσει. Είστε ιατρός ήδη, ε? είναι κάτι που προφανώ προφανώς είναι προσφυλέ. Ποιε είναι ε, οι εξελίξεις σχετικά. Και ένα-δυο λόγια και για τα εγκλήματα πολέμου. Βεβαίω και σα στηρίζουμε στην όλη προσπάθεια να πάυσει η ατιμορρησία για τα εγκλήματα πολέμου. Δεν θα πάρω μέρο για τα όσα ελέγχθησαν περί μεροληψίας, ποια από τις πλευρές πρέπει να υποστηριχθεί όχι, οι συνάδελφοι τα ξέρουν καλύτερα από μένα, αλλά λόγω του σεβασμού που έχουμε στη χώρα σας και στην, στον πολιτισμό σας, να σας πω απλώς ότι στην Ευρώπη παραμένουμε ενάντια στη θανατική ποινή. Ευχαριστούμε κυρία Νέιτς. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, εκ μέρους της αντιπροσωπείας μου και των φιλελευθέρων να σας καλωσορίσω. Ευχαριστούμε για την ομιλία σας σήμερα το πρωί εδώ. Η ομάδα μου ήταν μεταξύ των προτεργατών της κοινή λύση, του κοινού μάλλον για το Μπαγκλαντές. και κυρίως για τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα στον ε, τομέα της ένδυσης, στον βιομηχανία της ένδυσης χώρα τους περασμένους το είπαν και οι συνάδελφοι. Οι ευθύνε είναι κοινέ και τι επομίζονται πολύ διαφορετικοί φορεί και παράγοντε. Όχι μόνο οι αρχέ του Μπαγκλαντέ, αλλά και εμεί οι ίδιου καταναλωτέ και εν τέλει το σύστημα εποπτεία που διαθέτουμε που δεν παίρνει τα πράγματα αρκετά σοβαρά, δεν περνάει στην ουσία. Σας ενθαρρύνω λοιπόν και καλωσορίζω τις πρωτοβουλίες που προαναγγείλατε και θα ενθάρρυνα την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και τι αρχέ της χώρας να τις υλοποιήσουν. Είναι πολύ σημαντικό για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων του Μπαγκλαντέ να αναλυφθεί δράση. Μην ξεχνάμε ότι στους εργαζόμενους αυτούς η πλειονότητα είναι γυναίκες. Είναι σημαντικό αυτό λοιπόν και θα παρακολουθούμε τι προσπάθειε σα και με συμπάθεια και με διαρκή έλεγχο, ασκώντας διαρκή έλεγχο. Ως προς το δικαστήριο ε, που εξετάζει τα εγκλήματα τα οποία διαπράχθησαν κατά τον πόλεμο απελευθέρωσης και τις επακολούθες εμφύλιες συγκρούσεις, δεν ξέρω και εννοείται ότι δεν μπορούμε να διονύζουμε οποιαδήποτε μορφή ατιμορρησίας, όπως είπε ο συνάδελφος Ντεκεζέρ. Όλοι μας αισθανόμαστε και με κάθε τρόπο εναντιονόμαστε στη θανατική ποινή. Ελπίζαμε ότι θα είχε κρυζωθεί η θανατική ποινή σε όλη την Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες και θα ενθαρρύναμε κάθε χώρα στον κόσμο να κάνει ακριβώς το ίδιο. Κυρία Ντεμαρτίνη, ευχαριστώ ε, Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, σα ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα. Συγχαρητήρια για τα επιτεύγματά σα. Όχι μόνο για το 6% οικονομικής αύξησης ετησίω, αλλά επειδή μειώσατε την παιδική χρησιμότητα και τη βελτιώσατε την κατάσταση των ε, γυναικών, προωθώντα την έρευνα και την ε, παιδεία. Είμαι και εγώ ιατρό με σπουδέ στην Ιταλία και τι Ηνωμένες Πολιτείες στο Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς, πολύ κοντά Πρώτα ως φοιτήτρια και μετά ως καθηγήτρια. Έχουμε πολλά κοινά λοιπόν και έχω σπουδάσει και εγώ με τη σειρά μου πέρα από τις σπουδές μας μάλλον στο Λονδίνο. Για μένα θα είστε πάντοτε ένα πρότυπο για, τον, ε, για την δράση μου στο δημόσιο βίο. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mr. Chairman. A very warm welcome. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα θερμό καλωσόρισμα προ τον Υπουργό. Πρώτα απ' όλα, συλληπιτήρια στο λαό σα για την τραγική απώλεια ζωών μετά την κατάρρευση του εργοστασίου και του κτηρίου του. Είμαι ένας πραγματικός φίλος του Μπαγκλαντές, γιατί δεν θυμόμαστε συχνά ότι ένα εκατομμύριο ε, πολίτες του Μπαγκλαντές ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 100.000 μάλιστα είναι Βρετανοί. Και αυτό είναι για μας ένα πλεονέκτημα για την εκλογική μου περιφέρεια συγκεκριμένα, για το Λονδίνο. Έρχεστε λοιπόν από μια χώρα με πολύ ισχυρή παρουσία στις χώρες μας. Εγώ είμαι υπεύθυνο τη κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία που παρατήρησε τι πρόσφατε εκλογέ σα. Ήταν εντυπωσιακή η διεξαγωγή του με πολύ εύρυθμο τρόπο δεξίχθησαν όλα και ελπίζω αυτό να ε, επαναληφθεί και την επόμενη φορά. Για μένα ε, ε, είσαστε μια άξια εκπρόσωπο των Μπαγκλαντέ και του μεγάλου σεβασμού που δείχνει η χώρα σα για την εκπαίδευση των γυναικών ιδίω. Η πρωθυπουργό σα, εσεί ω υπουργό, η αρχηγό τη αντιπολίτευση και η εξαιρετική πρέσβη σας που, πρέσβυρα μάλλον που βρίσκεται στα δεξιά σα, σα το λε κυρίε με πολύ υψηλά προδιαγραφέ για τον δημόσιο βίο και μάλιστα δίνετε παράδειγμα για όλο τον κόσμο, ιδίω για τον Ισλαμικό. Πέρα από τον εγχώριο νόμο σας, το δίκαιο για, το, για τα εργατικά δικαιώματα, ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσει για τις ε, εκλογές στο Πακιστάν, γιατί είναι πολύ ισχυρές και αντίρροπες οι δυνάμεις ε, που έρχονται σε σύγκρουση στην πολιτική αρένα τις τελευταίες δεκαετίες, προερχόμενες και από την Ινδία πολλές φορές. Η Πρωθυπουργός θέλει χειρότερε θέσει με την Ινδία και η δική σα χώρα έχει και επιθυμεί στενότερε σχέσει με την Ινδία. Πώ βλέπετε να διαμορφώνεται το πολιτικό κλίμα για τι επόμενε εκλογέ μέσα ω Υπουργό Εξωτερικών. Και θέλετε να μα μιλήσετε και για, τη Ραχίγκα, ε, για το θέμα των Ραχίνγκα, των μουσουλμάνων Ραχίνγκα. Κάτι που επηρεάζει τι σχέσει σα ε, με την Βυρμανία ε, και την παρουσία των Ραχίνγκα εκεί πέρα. Ε, Επίση, να επαναλάβω και εγώ ότι τη τιμωρησία για τη γενοκτηνία δεν θα πρέπει να υπάρξει σε καμία περίπτωση. Επισκέφτηκα το Μουσείο των Εγκλημάτων Πολέμου, ε, γνωρίζω ποιοι ε, τη μνήμη διατηρείται από τους ήρωες του πολέμου της απελευθέρωσης και δεν ξεχνάω τις γυναίκες των εθνοτικών μειονοτήτων, Ινδουίστριες, Χριστιανές, Μουσουλμάνες που θα πρέπει να τις θυμόμαστε διαρκώς και Νομίζω απλώ πρέπει να ξεπεράσετε από το στάδιο τη ιστορία σα και να προχωρήσετε. Ήταν αποτρόπαια τα εγκλήματα που διαπράχθησαν τότε, αλλά σωστά έχετε αναλάβει δράση για να ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση. Ελπίζω ότι οι επόμενε εκλογέ σα θα είναι και ελεύθερε και δίκαιε και ότι θα πάει πολύ καλά η επόμενη επίσκεψή μα για την παρατήρηση των εκλογών. Και πάλι θερμό όρισμα και ευχαριστούμε για την ομιλία σα. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματικά κολακεύομαι από την καλοσύνη σας και από την ε, θερμή σας στήριξη προς τη χώρα μου και το λαό μου. Και προς την κυβέρνησή μου, αλλά και εμένα την ίδια. Σας ευχαριστώ θερμά. Η απάντησή μου στο ερώτημα για το αν είμαστε τακτικό μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας και αν έχουμε συνυπογράψει και κυρώσει τις σχετικές συμβάσεις. Ναι, είμαστε. Η νομοθεσία μας αντικατοπτρίζεται στις περισσότερε από τις υποχρεώσεις των συμβάσεων, απλώς με κάποια κενά. Διότι άρχισε να ισχύει ο νόμος από το 2006 μόλις και κατά το διάστημα εκείνο η Λίγκα Αουάμι, το δικό μου κόμμα, ήταν στην αντιπολίτευση. Και είχαμε προτείνει 54 τροπολογίες, των οποίων το σύνολο απορρίφθηκε από το κυβερνόν κόμμα. Έπρεπε μάλιστα να αποχωρήσουμε με τρόπο θεατρικό από το Κοινοβούλιο σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Έκτοτε, τις τροπολογίες αυτές τις συμπεριλάβουμε στο προεκλογικό μας ε, πρόγραμμα και έκτοτε ακούστηκαν φόβοι και γι' αυτό επιχειρήσαμε να διαμορφωθεί σύγκληση μεταξύ των ενδιαφερομένων. Προτείναμε λοιπόν τροπολογίε στο εργατικό δίκαιο, τον εργατικό μάλλον νόμο του 2006, νόμος ο οποίο έχει ήδη βελτιωθεί από την κυβέρνηση και θα αντικατασταθεί στην επόμενη ε, σύνοδο του Κοινοβουλίου που ξεκινά στι 3 Ιουνίου. Ελπίζουμε ότι οι τροπολογίες αυτές να περάσουν μέχρι το τέλο του Ιουνίου, να εγκριθούν. Και έτσι έχουμε την πεποίθηση καθώς είμαστε σε διαρκή επαφή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας, έχουμε την πεποίθηση ότι θα είμαστε πλέον σε θέση να καλύψουμε όλες τις ελλείψεις. Καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με βασικά θεμέλια, ε, τα πρώτα λιθαράκια της κατασκευής ενός τείχους ασφαλείας για όλους τους βιομηχανικούς κλάδους προστασίας δηλαδή των εργαζομένων. Για να απαντήσω και στο θέμα των υπεργολαβιών. Ναι, θα ασχοληθούμε και με το θέμα των πολλαπλών εξωτερικών συνεργατών, διότι, να είμαι εδώ ειλικρινής, μιλούμε για τη συμμόρφωση αλλά τι γίνεται με τους αγοραστές. Όταν πάνε να αγοράσουν τα προϊόντα μας, κοιτάνε λίγο, κάνουν μια έρευνα αγοράς και αγοράζουν τα φθηνότερα. Και κάποιες φορές, εν γνώση τους, κλείνουν τα μάτια στην ύπαρξη υπεργολαβιών. Ε, η κυβέρνηση κάνει το εξή αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο μάλιστα η κυβέρνηση, αλλά και η βιομηχανία μας και οι εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι ενδιαφερόμενοι και με στήριξη των ε, φίλων μας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ασχολούμαστε με όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί ακόμη και αν οι ε, είναι πολλοί, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις εργατικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις για την προστασία των εργαζομένων. Είναι τεράστιο καθήκον, αλλά με μεγάλη σημασία. Κοστίζει πολλά, αλλά πρέπει να γίνει και είμαστε απόλυτα ε, αποφασισμένοι να τα φέρουμε εις πέρας. Για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία και τη σχετική νομοθεσία, Υπάρχει μία ε, πρόταση για την εργασιακή ασφάλεια. Είναι θέμα εβδομάδων, ούτε καν μηνών το να περάσει. Μόλις λοιπόν περάσει και αυτός ο νόμος, με όλες τις πρωτοβουλίες που προβλέπει, και μόλις αρχίσουν να υλοποιούνται αυτές οι πρωτοβουλίες, νομίζω, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, ότι θα έχουμε αλλαγές και στην πράξη. Ορατές από όλους. Μέσα σε ένα χρόνο το πολύ υπολογίζω. Το θέμα της θανατικής ποινής. Το θέσατε πολλοί από εσά και καταλαβαίνουμε το την τοποθέτησή σα. Γνωρίζουμε καλά τη θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη θανατική ποινή. Όμως ενώ σεβόμαστε αυτήν την γραμμή, να πω ότι δεν υπάρχει συνολικά συνένεση για το τι θα απογίνει με τη θανατική ποινή. Σε πολλά μέρη του κόσμου παραμένει, ακόμη και σε κάποιες δυτικές χώρες ισχύει και επιβάλλεται η θανατική ποινή. Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει στο πλαίσιο της αναθεώρησης του συνολικού, του συνολικού συστήματος ποινικού δικαίου, δεδομένων μάλιστα και των οικονομικών συνθήκων του Μπαγκλαντές, έτσι κι η ποινή αυτή επιβάλλεται σε περίπτωση πραγματικά φρικτών εγκλημάτων. Δεν ανατρέχουμε σε αυτήν συχνά. Μόνο σε περιπτώσεις φρικτών, ε, αποτρόπαιων εγκλημάτων. Ε, μέχρι να αποφασιστεί μάλιστα η επιβολή τη, γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι, πάρα πολλέ ε, δοκιμέ και πραγματικά είναι σπανιότατε περιπτώσει όπου χρησιμοποιείται. Θα θέλαμε λοιπόν εδώ την ανοχή και την κατανόησή σα. Είναι μέρο του νομικού μα συστήματο. Και πρέπει βεβαίω, εκμεταλλευόμενοι αυτή την ευκαιρία, να μοιραστώ και το εξή μαζί σα. Ένα από τα πιο πρόσφατα φαινόμενα στο Μπαγκλαντές. Από το Διεθνές Δικαστήριο για τα Εγκλήματα Πολέμου επιβλήθηκε διαβίου κάθριξη ισόβια σε έναν από τους εγκληματίες πολέμου. Ξαφνικά λοιπόν ε, κινητοποιήθηκε ολόκληρη η νεολαία της χώρας με εκατοντάδες χιλιάδες νέους στους δρόμους. Συγκεντρώσεις στο κέντρο των πόλεων. Αυτό ονομάστηκε το κίνημα Σάμπαρ. Συγκεντρώνονταν και έμεναν στους δρόμους επί ένα δίμηνο, ξανά και ξανά, μέχρι πρόσφατα. Δεν μένουν όλο το 24 φυσικά στο ίδιο σημείο, αλλά πάνε και έρχονται και οργανώνουν τη διαμαρτυρία τους κατά αυτόν τον τρόπο. Διαμαρτύρονταν και έλεγαν οι νέοι γιατί, ρωτούσαν γιατί κάποιος που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη σκότωσε 350 ανθρώπους και έκανε, διέπραξε και άλλα εγκλήματα. Γιατί λοιπόν καταδικαστεί απλώ σε ισόβια κάθεξη. Πόσου έπρεπε να έχει σκοτώσει για να πάρει τη θανατική ποινή, για να του επιβληθεί η θανατική ποινή. Σα μιλάω για κίνημα νεολαία. Ολόκληρη χώρα κινητοποιήθηκε. Το μεγαλύτερο μέρο των πολιτών είναι μαζί του. Έτσι τοποθετεί. Αυτό είναι το κοινό αίσθημα. Σα ζητώ λοιπόν να καταλάβετε πώ αισθάνονται και τα θύματα των όσων έγιναν το 1971 και οι οικογένειές τους, είτε 300.000 γυναίκες που βασανίστηκαν και διάστηκαν το 1971 και 3 εκατομμύρια άνθρωποι που θανατώθηκαν, δολοφονήθηκαν. Μιλάμε για μια βαθιά πληγή, ένα τραύμα που έχει παραμείνει ανοιχτό στη χώρα μας για τα τελευταία 42 χρόνια. Προσπαθείτε να το δείτε και από αυτή τη σκοπιά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Τσάρλς, για την εξωτερική μας πολιτική και ως προς τις σχέσεις μας με την Ινδία και το Πακιστάν. καλωσορίζουμε την χειρονομία των ε, κλεγέντος Πρωθυπουργού του Πακιστάν, του κυρίου Σαρίφ, διότι αυτή η κίνηση προ την Ινδία, καθώ και η θερμή απόκριση τη Ινδία είναι θετικά δείγματα. Πιστεύουμε ότι στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή μα πρέπει να υπάρξει ειρήνη. Ειρήνη, ασφάλεια και ανάπτυξη. Ο Πρωθυπουργό μα, ή Πρωθυπουργό μα, όταν ανέλαβε καθήκοντα για δεύτερη φορά, δεύτερη φορά στις αρχές του Ιανουαρίου του 2009, απίφθινε έκκληση προς όλες τις όμορες χώρες και τις γείτονες χώρες να συνεργαστούμε λέγοντας ότι έχουμε έναν κοινό εχθρό, έναν, την ένδια, τη φτώχεια και ότι θα πρέπει πάντοτε να ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να ξεφεύγουμε από αυτή την απειλή που ελοχεύει. Πρέπει να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε μια καλύτερη ζωή σε όλους μας τους ε, ανθρώπους στο λαό, στους λαούς μας που αξίζουν πολύ περισσότερα. Αυτό επιδιώκουμε και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Μπορώ να σας πω με σχετική περηφάνεια ότι χάρη τις ε, ε, αδιάκοπες προσπάθειες της Πρωθυπουργού μας και την επιμονή της, έχουμε πλέον στην Νοτιοανατολική Ασία ένα τέτοιο κλίμα που επιτρέπει τη συνεργασία, την συνεργασία προς την επίτευξη κοινών στόχων, για να ξεφύγουμε ακριβώς από την απειλή της στόχιας. Δημιουργήθηκε ένα κλίμα συνεργασίας ε, και διαλόγου αντί για την εχθρότητα που υπήρχε στο παρελθόν. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, το Μπαγκλαντές θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον ίδιο ρόλο σε αυτήν την ε, γεωγραφική ζώνη, ώστε να δημιουργεί συνθήκες που νευνονούν την ειρήνη, να την προστατεύει και να οδεύει προς την δημοκρατία, την ενδυνάμωσή της, την ενδυνάμωση των θεσμών και προστατεύοντας τα δικαιώματα των ανθρώπων σε κάθε δυνατό επίπεδο. Για το θέμα των Ροχίνγκα, των μουσουλμάνων Ροχίνγκα, είναι δυστυχώ μια τυχή περίπτωση. Οι Ροχίνγκα έχουν γίνει ένα πρόβλημα που διονύζεται εδώ και τρεις δεκαετίες. Το Μπαγκλαντές Εξαιτία και τη πείρας που είχε, της εμπειρίας που είχε το 1971, όταν 10 εκατομμύρια πολιτών μας έγιναν πρόσφυγε σε διαφορετικά γειτονικά κράτη, στην Ινδία κυρίω. Ακριβώ για αυτόν τον λόγο προσπαθούσαμε και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για του ανθρώπου αυτού. Για του Ροχίνγκα που ε, δραπετεύουν από τη Βυρμανία, από το Μιανμάρ και προσπαθούν να γλιτώσουν από βασανιστήρια και διώξει. Είμαστε όσο καλύτεροι οικοδεσπότε γίνεται. Έχουμε περίπου 29.000 πρόσφυγε αυτή τη στιγμή, επισήμω καταγεγραμμένου σε δύο καταβλισμού προσφύγων. Εκεί, με τη βοήθεια της ΥΠΑ της Αρμοπιστία του ΟΗΕ και κάποιων φίλων μας, τους φροντίζουμε όσο μπορούμε. Όμως, υπάρχουν ακόμα 300-500 χιλιάδες παράνομοι, τέλος πάντων χωρίς επίσημα χαρτιά ροχίνγκα που έχουν μπει στην επικρατειά μας. Και αυτό είναι τεράστιο άρθρος για μια χώρα η οποία είναι από τις πολυπληθέστερες, από τις πιο πυκνοκατοικημένες μάλλον στον κόσμο. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλους. Πρακτικά είναι αδύνατο να δεχτούμε άλλους πρόσφυγες. Γι' αυτό σας το λέω ξεκάθαρα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλους. Το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Σε διμερή βάση διαπραγματευόμαστε με το Μιανμάρ για τον επαναπατρισμό αυτών των Ροχίγκα. Δεν έχουμε κυρώσει την ε, Σύμβαση για τους Πρόσφυγες, ούτε τα πρωτοκολλά της. Διατηρούμε την πολιτική της μη επαναπρόθεσης και ουδέποτε ξαναστήλαμε πίσω κανέναν με το ζόρι, με τη βία, αλλά δεν αντέχουμε άλλο. Δυστυχώς αυτή είναι τώρα η θέση μας και είναι πραγματικά τεράστιο το βάρος ούτε περιβαλλοντικά, ούτε οικονομικά, ούτε από την άποψη του κράτους δικαίου και της στήριξη της τάξης μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Κάποια από τους Ροχίγκα που κάποιες φορές διέρχονται απλώς από τον Παγκαντές για να φτάσουν ε, σε άλλα κράτη, δημιουργούν προβλήματα και στην αγορά εργασία. Κλέβουν δουλειές από τους ε, πολίτες του Μπαγκλαντές. Επηρεάζουν την ε, δουλειά, τις δουλειές στη χώρα μας και καταστρέφουν και την εικόνα των εργαζομένων μας που κατά τα άλλα είναι γνωστοί ως ε, πολύ πειθαρχημένοι, σκληρά εργαζόμενοι, ευσυνείδητοι εργαζόμενοι. Και αυτό σε πολλές διαφορετικές χώρες. Είναι λοιπόν ένα πραγματικό πρόβλημα για μας και ελπίζουμε ότι όλοι θα μας βοηθήσουν. Το Μιανμάρ, ε, θα βοηθήσουν μάλλον το Μιανμάρ για να βρεθεί λύση. Το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί και εκεί πρέπει να βρεθεί λύση. Είναι θέμα των δικαιωμάτων που δίνει το Μιαμάρ στους πολίτες της και ε, πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιες οικονομικές συνθήκες, ένα περιβάλλον ευνοϊκό, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορέσουν να επιστρέψουν στο Μιαμάρ και να αισθάνονται ε, ασφαλείς στην πατρίδα τους. Συνεργαζόμαστε με τους γειτονές μας και απευθείας με τις Βρυμανικές αρχές, το Μιανμάρ, για να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Ελπίζουμε και εδώ να δείξετε κατανόηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν όλους σας που είστε στο πλευρό μας. Σε αυτές τις στιγμές, ε, αμέσως μετά την ε, μεγάλη αυτή τραγωδία που έτυχε. Ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε και δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και περνάει από το χέρι μας για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Όμως υπάρχουν κατά πάσα πιθανότητα ακόμα πολλά κτίρια που δεν είναι ασφαλή διότι αυτό είναι έκφανση της ατιμορρησίας που επικρατούσε στη χώρα επί δεκαετίες όταν οι άνθρωποι διέπραταν γενοκτονίες, δολοφονούσαν τον πατέρα του έθνους και σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαμε το μυαλό τότε να σκεφτούμε ότι τα κτίρια μας δεν ήταν αρκετά ασφαλή και δεν σέβονται τις προδιαγραφές ασφαλείας. Ατιμορρησία λοιπόν την οποία προσπαθούμε να εξαλείψουμε. Σε αυτό το ταξίδι ελπίζουμε ότι θα σας έχουμε συνοδοιπόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο. Σας θέλουμε στο πλευρό μας. Όπως συνέβαινε ανέκαθεν. Σας ευχαριστώ πραγματικά θερμά για τη στήριξή σα. Ευχαριστώ. Thank you very much, Minister. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ, για τις πληροφορίες σας και την προθυμία να συζητήσετε επίσης μαζί μας αυτά τα τραγικά γεγονότα. I hope... Και ελπίζω ότι θα αποφύγουμε κάτι τέτοιο στο μέλλον. Δεν είναι μόνο δουλειά της χώρας σας. Συζητούμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα θέματα. Επειδή οι δικές μας εταιρείες που προσπαθούν φθηνά εμπορεύματα να διαθέσουν στην Ευρώπη και οι εταιρείε μας είναι υπεύθυνε. Πρέπει να καταστήσουμε λοιπόν σαφές ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείε πουλώντας τέτοια φθηνά προϊόντα στην Ευρώπη πρέπει να εφαρμόσουν κάποιους συγκεκριμένους κανόνες προστασίας των εργαζομένων, των εργατών εκεί και κοινωνικές προδιαγραφές και της ε, ίδιας της αγοράς του Διεθνούς Γραφείου Οργανισμού Εργασίας ε, ώστε να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και ελπίζω ότι από κοινού θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν θέση απασχόλησης, θέση εργασίας αλλά με αξιοπρεπείς μισθούς και καλύτερους όρους απασχόλησης. Δεν πρέπει να εκμεταλλεύεται η Ευρώπη θα έλεγα την κατάσταση, μια κακή κατάσταση επιτόπου κάποιων χωρών όπως ε, τις συνθήκε στη χώρα σας. Και είναι λοιπόν κοινή μας ευθύνη να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ Υπουργέ. Thank that is written by our father. Και τώρα περνάμε στην πραγματικά, στο επιστέγασμα της uh, τριμερούς συνεδρίασής μας, την έκθεση του κύριου Κούκαν. Παρακαλώ, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Με πολύ ωραίο κομψό τρόπο το είπατε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, στις 29 και 30 Απριλίου είχαμε την έκτη συνάντηση σταθεροποιητικής επιτροπής και σύνδεσης ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγινε, έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου Ποντγκόριτσα. Έξι μέλη σε σχέση με την αντιπροσωπεία μας. Γιέλκο Κάτσιν, Άννα Ιμπρισάγκητς, Φραντσέσκο Ντε Άντζελες Νίκος Χρυσόγελος και Ουλρίκε Λούνατσεκ και εγώ είχαμε δύο συνεδριάσεις με τους συναδέλφους μας ε, του Κοινοβουλίου και πριν συναντήσαμε τους πολιτικούς ηγέτες της χώρας, τον πρόεδρο, πρωθυπουργό και δύο αναπληρωτές υπουργούς. Η αντιπροσωπεία μας ήταν η πρώτη υψηλού επίπεδου αντιπροσωπεία που πήγε εκεί μετά από τις εκλογές που ήταν επίμαχες ως προς το αποτέλεσμα. Όταν όμως εμείς πήγαμε εκεί είχαν τελεσιδικήσει τα αποτελέσματα των εκλογών. Επισκεφθήκαμε με, κατά τη διάρκεια μιας, ε, ενός μποϊκότ του Κοινοβουλίου τρία από έξι αντιπολιτευόμενα κόμματα ε, μποϊκόταραν το κοινοβούλιο. Το θέμα των εκλογών ήταν ένα θέμα κλειδί για, αυτές, ε, για αυτή την κατάσταση και η συζήτηση για το σκάνδαλο των ε, οπτικοακουστικών μαγνητοσκοπήσεων και καταλήξαμε σε αυτό το μποϊκό του Κοινοβουλίου. Αυτό επισκίασε τα θέματα σε σχέση με την μάχη των αγώνα κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου ε, εγκλήματος. Δύο λόγια για την ενημέρωσή σας. Πρόσφατα είχαμε την διαρροή για τέτοιου είδους μαγνητοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκε αναφέρθηκε πώς, μπορούσαν να πώς χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά κονδύλια και από χορηγίες προς όφελος των γνωστών ε, εκείνων ε, οπαδών ε, κόμματος. Αυτό το κόμμα ήταν πραγματικά κάτι, αυτό, αυτή η διαρροή και αυτό το σκάνδαλο υπονόμευσε τα πράγματα και συνέπεσε με τις προ, προεδρικές εκλογές του Απριλίου επηρεάζοντάς, τα σοβαρά και είχαμε μια πολύ μικρή πλειοψηφία και τα αποτελέσματα ακόμα δεν αναγνωρίζονται μέχρι σήμερα από την αντιπολίτευση. Και υπό αυτούς τους όρους πήγε η αντιπροσωπεία μας εκεί. Και μπορεί κανείς να συνοψίσει τα πράγματα ως εξή. Το σκάνδαλο το οπτικοακουστικό πρέπει να, τύχει πολιτικής, να έχει πολιτική συνέχεια και δικαστική συνέχεια και θα πρέπει να κριθούν τα πράγματα μέσω των κριτηρίων της Κοπενχάγης. Τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών είναι τελικά πλέον και δεν πρόκειται να συζητηθούν. Οι ελλείψεις του εκλογικού συστήματος είναι σοβαρές και εξακολουθούν να υφίστανται από τη μία εκλογή στην επόμενη. Πρέπει να βελτιωθεί αυτό το εκλογικό σύστημα στο Μαυροβούνιο πριν από τις επόμενες εκλογές οι ανησυχίες και τα μελήματα της αντιπολίτευσης εν μέρη δικαιολογούνται και πρέπει να αντιμετωπιστούν και να διευθετηθούν από τις αρχές. Παρότι όμως το κύριο αίτημα αναφέρεται ότι δεν είναι συνταγματικό, δηλαδή το μποϊκοτάρισμα του Κοινοβουλίου δεν μπορεί να υποστηριχθεί υπό κανένα όρο και προϋπόθεση και σε σχέση με τα προβλήματα αυτά αν δεν αντιμετωπιστούν με το σωστό τρόπο και δεν υπάρξει, δεν εμφυσιθεί ε, εμπιστοσύνη στις ε, δημοκρατικές διαδικασίες και δεν αποκατασταθεί το δημοκρατικό κύρος θα υπονομευθεί η κατάσταση στο Μαυροβούνιο. Έτσι παρουσιάστηκαν τα πράγματα και στο Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου και έτσι και στις διπλωματικές επαφές παρουσιάστηκαν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο πρόεδρος ε, του Κοινοβουλίου προσπαθεί να βρει τρόπο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να βελτιωθούν τα πράγματα. Φαίνεται ότι ανταποκρίνεται στα αιτήματα της αντιπολίτευσης καθώς όλα αυτά είναι συνταγματικού χαρακτήρα. Όμως ταυτόχρονα εν μέρει αναγνωρίζει τα προβλήματα η κυβέρνηση. Υπόσχεται όμως ε, να τα αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά με τον ορθότερο τρόπο. Ένα κοινό έγγραφο υιοθετήθηκε κατά το τέλος της συνεδρίασης, έχει και παραγράφους ε, για τις προεδρικές εκλογές που συμπεριλαμβάνει εν συνόψη, εν περιλήψη, ανησυχεί το κοινό, οι πολίτες ε, για το σκάνδαλο αυτό των οπτικοακουστικών αυτών ε, μέσων και τις ε, παρατυπίες. Υπάρχει πολιτική, πολιτικό ζήτημα εδώ και με πολύ μεγάλη προσοχή εξετάστηκε το θέμα αυτό στο Μαυροβούνιο. Η αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου παρουσίασε μια ενιαία και συνεκτική θέση που έγινε δεκτή με κατανόηση από όλες τις πλευρές. Οι συζητήσεις για την εξουσία στο Μαυροβούνιο αφορούν πολλά άλλα θέματα, όμως ελπίζω ότι θα ήταν σκόπιμο μόνο τα ουσιοδέστερα να αναφερθούν. Και θέλω να προσθέσω ότι κατά τη διάρκεια αυτής της ε, τρίτης ε, είχαμε και τον ε, Υπουργό Εξωτερικών και τον κύριο Λούξιτς και τη συνάντηση του διαβριμένου προεδρίου μας ενημέρωσε ότι αυτή την εβδομάδα, σήμερα ακριβώς, θα υπάρχει μια έκτακτη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου και θα ήθελα να παρουσιάσουν την λύση πώς να αντιμετωπιστούν τα αιτήματα της αντιπολίτευσης, είπε και αναμένει να επιτευχθεί συμφωνία για την επίλυση και διαθέτηση της κατάστασης και να πάψει το μποϊκό του Κοινοβουλίου, το μποϊκοτάρισμα του Κοινοβουλίου με αυτόν τον τρόπο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, Πρόεδρε. Τάνοκ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σύντομα, να πω πως εγώ εμπιστεύομαι πλήρως τον Εντουαρτ Κούκαν, είναι ο βασικότερος ε, ειδικό για τα Βαλκάνια στην Επιτροπή μας, πρώην υπουργό Εξωτερικών, διπλωμάτης, οπότε ο συγητής δεν μπορώ να αμφισβητήσω οτιδήποτε. Δεν ήμουν παρόν στις εκλογές, ε, διάβασα μόνο τα σχετικά. Χαίρομαι για το ότι η κατάσταση ομαλοποιήθηκε, θα αντληθούν διδάγματα από την εμπειρία αυτή όσον αφορά τα ελλείμματα στην εκλογική διαδικασία. Προφανώς ε, ο πρόεδρος έχει ελάχιστες εκτελεστικές εξουσίες και είναι ένα συμβολικό αξίωμα, είναι πρωθυπουργικό το σύστημα και κοινοβουλευτικό, οπότε προφανώς οποιαδήποτε παρατυπία πρέπει να διερευνηθεί, αλλά νομίζω συνολικά όλα τα κόμματα δέχονται το αποτέλεσμα και το Κοινοβούλιο θα ε, επαναλάβει τις εργασίες του θα σταματήσει τον μποϊκοτάζ από την αντιπολίτευση. Ήμουν παρόν και σε μια συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Λούξικ που μας διαβεβαίωσε πως τα πράγματα θα επιστρέψουν στην ομαλότητα σύντομα. Το Μαυροβούνιο είναι μικρή χώρα, όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους. Μικρή, σφιχτή κοινωνία, ευημερή. Είναι αυτή τη στιγμή η μόνη χώρα που διαπραγματεύεται στα Δυτικά Βαλκάνια για ένταξη. Πρέπει να την στηρίξουμε. Ελπίζω να έχει λήξει τώρα το ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο, ο πρόεδρος. Θέλετε να απαντήσετε. Δεν ε, έκανα κάποια ερώτηση. Καμιά φορά μπορεί να με... Δεν ξέρω, μπορεί να μην του άρεσε η δήλωσή σας, λέει ο πρόεδρος. Συμβαίνουν και αυτά. έλαβα την δήλωση του κυρίου Τάνοκ, ε, την άκουσα μάλλον, με συγχωρείτε, ε, πάρα πολύ θετική. Μάλιστα, τι σημειώνετε. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λύεται η συνεδρίαση. 12 o'clock, η ώρα, σε 5 λεπτά διευρυμένο προεδρείο.